Μένα το κύριο που είναι εδώ, την κυρία Ράπτη, σας ανέφερα πρώτη, πρώτη κυρία Ράπτη και κατόπιν ε, θα δώσω το λόγο και στους υπολείπους ε, και να καλωσορίσω και τον κύριο Κρός, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, της Διεύθυνσης ΓΔΕΛΤΑ Έρευνας και Ανάπτυξης. Κυρία Κόμη, ευχαρίστω να σας δώσω το λόγο καταρχήν για να παρουσιάσετε τη γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν να παρουσιάσω το κείμενο αυτής της γνωμοδότησης, θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Καταρχήν, το θέμα είναι πολύ ευρύ και ενδιαφέρον. Πρόκειται για ένα από τους πιο σημαντικούς ε, φακέλους που έχουμε σε αυτή τη θητεία. Ήθελα να προσθέσω και κάποιες λεπτομέρειες για ορισμένα σημεία που έχω συμπεριλάβει στο κείμενο και κάποια άλλα στοιχεία σε σχέση με σημαντικές ε, πτυχές. Αλλά έπρεπε να σεβαστώ το όριο των χαρακτήρων. Για το λόγο αυτό εκπονώ μια σειρά πρόσθετων τροπολογιών που θα συμπληρώσουν το κείμενο και αν κάποιο από εσά ενδιαφέρεται ε, μπορεί φυσικά να έρθει σε επαφή με το γραφείο μου γιατί θεωρώ ότι αυτή η Επιτροπή πολύ συγκεκριμένα ιστορικής αγοράς ε, έχει συγκεκριμένη σχέση και με το Single Market Act και λειτουργεί στρατηγικά στο ιστορικό αυτού του φακέλου. Για να περάσω στην ουσία της υπόθεσης ε, θεώρησα ότι είναι ουσιαστικό να ζητήσω συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων Έρευνα και κοινοτομία και των ταμείων συνοχή μέσω μία ενίσχυση των ρόλων της τοπικής αυτοδιοίκησης γιατί ε, σίγουρα θα έχουμε ε, ένα πέρασμα από ε, ένα ρόλο που διαδραματίζεται σε εθνικό επίπεδο σε ένα ρόλο που διαδραματίζουν οι ίδιες οι περιφέρειες. Ένα άλλο σχετικό θέμα έχει να κάνει με την απλούστευση των διαδικασιών μέσω της εισαγωγής μηχανισμών όπως είναι η σιωπηρή συνένεση και ε, ε, αυτό για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στα σχέδια και σε διάφορες πρωτοβουλίες όπως το χάρη τις κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες JITs για να, να υιοθετηθούν προγράμματα ευελιξίας είναι επίσης πολύ σημαντικό ε, για να μπορέσουμε να σεβαστούμε και την ταχύτητα των παγκοσμίων αλλαγών θα είναι λοιπόν απαραίτητο να προσπαθήσουμε να έχουμε συνεχές feedback ε, και σε ενδιάμεσο στάδιο αυτού του προγράμματος πλαίσιο σε ό,τι αφορά ελλαγέ, νέες τεχνολογίες και έρευνα θα πρέπει πάντοτε να συμβαδίζουν με το πέρασμα του χρόνου και μάλιστα να λαμβάνω την υπόψη και οι ανάγκε των πολιτών. Πιστεύω επίση ότι είναι απαραίτητο να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ενώ τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, ένα ποσοστό ε, του προϋπολογισμού για την έρευνα για να δημιουργηθούν κλάστερ. Εγώ θεωρώ ότι τα κλάστερ ε, δεν θα πρέπει να αποτελούνται μόνο και αποκλειστικά από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά θα πρέπει να αποτελούν ένα συνεχή τομέα δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται εκεί και τα πανεπιστήμια και μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να υπάρχει μια εγκάρσια εμπλοκή και συμμετοχή έτσι λοιπόν αυτό το προωθούμε και όχι μόνο σε περιφερειακό, συγγνώμη, σε εδαφικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή, να λάβουμε υπόψη, θέλουμε τις διάφορες ευρωπαϊκές πραγματικότητε. Η Κομισιόν θα πρέπει να δοκιμάσει και νέου τρόπους χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων εγώ προτείνω το βάουτσερ για την καινοτομία. Δεν μπόρεσα να το εξηγήσω λεπτομερώ στη γνωμοδότησή μου, αλλά θα ε, τύχει τροπολογία. Αυτό είναι ένα μέσο βεβαίως καινοτόμο, ένα νέο μέσο το οποίο θα επιτρέψει να δοθούν σε όλους η δυνατότητα να καινοτομήσουν. Ε, και μάλιστα και με μηδενικό κόστος σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, στο κοινό πλαίσιο θέλουμε να αξιολογήσουμε ένα πειραματισμό που θα βασίζεται στην αρχή της χρηματοδότησης με το βάουτσερ προκειμένου οι επιχειρήσεις να έρθουν πιο κοντά στα θέματα της καινοτομία και της ανάπτυξης χρησιμοποιώντας ένα σύστημα όπου διάφοροι όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες ο μηχανισμό θα μπορούσε να προβλέψει ε, να υπάρχει χρηματοδότηση μέσω αυτού του βάουτσερ. Προβλέπεται η χρηματοδότηση επιχειρήσεων που αποδεικνύουν ε, ότι ε, μπορεί να έχουν κάποιες εφαρμογές ή καινοτόμες προτάσεις τους και να χρηματοδοτούνται μέσω του βάουτσερ. Στην περίπτωση αυτή τα βάουτσερ θα είχαν ως στόχο να είναι, και συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτό τον όρο, ναι, ναι, να μιλήσω πιο αργά, λέει ο μιλήτρια. Έτσι λοιπόν ε, θα είχαν το στόχο να θεωρούνται ως κάποιες καλές δαπάνες, αν μπορούμε να το πλουστεύσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ότι δίνονται στις επιχειρήσεις που θέλουν να καινοτομήσουν και στη συνέχεια δαπανώνται ε, σε κάποια κέντρα. Έχουμε κάποια κέντρα ε, αριστείας όπω το JRC, ε, το Joint Research Center. Πολλέ φορέ δεν χρησιμοποιείται παρκώ από τι μικρέ και μεσέ επιχειρήσει. Έτσι λοιπόν αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο χρησιμεύει για να υπάρχει περιττέρω διευκόλυνση. Έτσι λοιπόν δεν θα πρέπει... Ε, μάλλον ουσιαστικά η χρήση αυτών των βάουτσερ θα πιστοποιείται από τα ίδια τα κέντρα έρευνα, τα οποία θα δαπανάτε το βάουτσερ. Έτσι λοιπόν αυτό θα σήμαινε δραστική απλούστευση των διαδικασιών και θα αποτελούσε ε, ένα καινοτόμο τρόπο και ένα επικορικό τρόπο για να υποστηρίξουμε τις ε, καινούργιες και καινοτόμες ε, πραγματικότητες. Θα μπορούσαμε να έχουμε είτε ε, περιφερειακή είτε εθνική χρηματοδότηση με την έγκριση ενός ευρωπαϊκού οργανισμού, δηλαδή μέσω μιας ευρωπαϊκής δομής η οποία θα επικύρωνε τη χρηματοδότηση αυτών των κέντρων. Αυτό ισχύει κυρίως για το JRC. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του και θα πρέπει να ε, συνεργαστεί περαιτέρω με τον επιχειρηματικό κόσμο. Αφιερώνω σε αυτό συγκεκριμένο σημείο. Τέλο. Άλλε πτυχέ επίση σημαντικές είναι η εισαγωγή της υπεροχής ε, των ε, κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, venture capital και ε, των εξοκοινοτικών επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στα project γιατί και αυτές μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στις έρευνές μας αλλά φυσικά θα πρέπει να υπόκεινται σε έναν ευρωπαϊκό συντονισμό θα εισαγάγω και κάποιο σημείο που δεν μου επιτρέπει γιατί δεν υπήρχε επαρκές χώρος στο σχέδιο γνωμοδότησης που θα αφορά το θέμα της ενίσχυσης της τυποποίησης και του συντονισμού με τα ερευνητικά προγράμματα. Χρειάζεται να υπάρχουν προτεραιότητες ε, σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και όχι πλέον σε συγκεκριμένο εθνικό επίπεδο και ο ρόλο των διαγωνισμών και τη πνευματική ιδιοκτησία των σχετικών δικαιωμάτων. Γιατί πολλέ φορέ Έχουμε εξαιρετική έρευνα, αλλά δεν προστατεύονται οι έρευνες αυτές με τον κατάλληλο τρόπο. Έτσι λοιπόν, ε, ουσιαστικά ε, δεν έχουμε και την ορθή μελλοντική εφαρμογή ε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε πρόταση, τροπολογία ή για ε, οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορεί να επιθυμείτε σε σχέση με όλα όσα έχω συμπεριλάβει στο σχέδιο γνωμοδότησης. Θεωρώ ότι η δική μας γνωμοδότηση ε, είναι μια γνωμοδότηση στο εσωτερικό της Επιτροπής Ήτρε, αλλά ίσως θα πρέπει να αποτελεί κάτι περαιτέρω από μια κατεύθυνση ε, που δίνει η εσωτερική αγορά σε αυτό το πρόγραμμα έρευνα. Γιατί αν θέλουμε να θέσουμε σε εφαρμογή την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς η έρευνα και η καινοτομία είναι οι λέξεις κλειδιά επί των οποίων θα πρέπει να εργαστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα αναλυτικά μας είπατε για την ε, έκθεση. Θα ξεκινήσει σύντομα η, έκθεση, η συζήτηση των σκιωδών. Πριν γίνει αυτό, να καλωσορίσω έναν απληρωματικό μέλος της Επιτροπής μας, την κυρία Γκάλο που ήρθε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κάνει πολύ καλή δουλειά στην ε, πνευματική ιδιοκτησία και αναμένουμε βεβαίω και τη συνεργασία, μας, συνεργασία σας μαζί μας. Αναμένουμε τώρα τις παρεμβάσεις των σκιωδών, ξεκινώντας από την κυρία Ράπτη. Κύριε Πρόεδρε, ακούγομαι, ναι. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ την κυρία Κόμη για το πολύ καλό κείμενο βάσης. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα καλό κείμενο πάνω στο οποίο να εργαστούμε. Ε, από το κείμενο αυτό στέκομαι ιδιαίτερα στην ενίσχυση της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ένα σημείο που εκτιμώ πάρα πολύ, μου αρέσει πολύ, θεωρώ ότι είναι το μέλλον για την Ευρώπη. Ε, μου άρεσε επίσης το θέμα της ε, σύμπραξης ε, ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων στο θέμα της καινοτομίας και της έρευνας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Κατανοώ επίσης ότι θα ήθελε πάρα πολλά άλλα πράγματα να περιλάβει και λόγω του γνωστού προβλήματος, εγώ το λέω πρόβλημα, δεν το λέω κανόνα, του να έχουμε μόνο μία σελίδα και συγκεκριμένες λέξεις, δεν μπόρεσε να βάλει όλα αυτά που πολύ θα ήθελε. Σκέπτομαι λοιπόν ότι προφανώς ανάμεσα σε αυτά που θα θα ήθελε να περιλάβει είναι μερικά πράγματα που σκέπτομαι κι εγώ. Ε, ξεκινώ λοιπόν και λέω θεωρώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να τονίσουμε το θέμα της διαφάνειας ε, βλέπω στο σημείο 3 της πρότασης που γίνεται αναφορά στο σημείο της σιωπηρής συνένεσης και σε εξαίρεση κατά κατηγορία. Ε, θα ήθελα να ακούσω κάποια περισσότερα πράγματα γιατί αυτά τα δύο σημεία ε, συν το σημείο των vouchers, των κουπονιών, νομίζω ότι πρέπει, είναι πολύ καλή πρωτοβουλία, πολύ καλή ιδέα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν κοντά τους και το θέμα της διαφάνειας και του ελέγχου. Υπάρχει επίσης το θέμα της ενημέρωσης που θα πρέπει να, για το οποίο θα πρέπει να λάβουμε πρόνοια, ε, ώστε οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες να ξέρουν πού υπάρχουν όλα αυτά τα καινοτόμα προϊόντα που μπορούν να τα, να τα χρησιμοποιήσουν. Και τελειώνω λέγοντας ότι ε, έχω την αίσθηση πως θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση και την κοινωνική διάσταση της εσωτερικής αγοράς θυμάμαι πάντα κάθε φορά που κουβεντιάζουμε ε, σε αυτή εδώ την επιτροπή για, για τον ανταγωνισμό για την εσωτερική αγορά θυμάμαι πάντα την έκθεση του κυρίου μόντι. θυμάμαι εκείνο το σημείο που ανέφερε στις πρώτες σελίδες ότι αυτή η εσωτερική αγορά δεν είναι ελκυστική και μονίμως σκέπτομαι ότι πρέπει να την κάνουμε ελκυστική και ένας τρόπος για να την κάνουμε ελκυστική είναι να πιστέψουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αυτό που πραγματικά πιστεύω ότι όλοι μας θέλουμε να κάνουμε, ότι θέλουμε να τους φροντίσουμε ε, θα ήθελα λοιπόν και αυτό το σημείο να το δω μέσα σε αυτή την έκθεση και βέβαια είμαι στη διάθεση της εισηγήτριας εάν μπορούμε να κάνουμε οποιασδήποτε ε, και τροπολογίες που και εγώ έχω στο μυαλό μου και άλλοι συνάδελφοι και αν μπορούσαμε ενδεχομένω και κοινέ τροπολογίες σε αυτές τις κατευθύνσεις που προανέφερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για τη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Μπουζόη. Ναι. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λερκόμη για το πολυθετικό ε, που σχέδιο κειμένου που μας παρουσίασε σήμερα. Επιμένουμε στην κοινοτομία και στην έρευνα. Είναι η στιγμή να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες λύσεις για να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό το τομέα, συνεισφέροντας έτσι στη μελλοντική μας ε, οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχει σημαντικός αριθμός ενδιαφέρουσων ιδεών που θα ήθελα να υποστηρίξω, όπως ο συντονισμός μεταξύ ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων καινοτομία ε, που θα υποστηρίζουν τα δίκτυα αριστείας και τα κλάστερ και για την ανάπτυξη ΣΔΙΤ ή τη συμμετοχή κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε προγράμματα έρευνα και καινοτομία. Ξέρω ότι υπάρχει ένα περιορισμό χαρακτήρων στο σχέδιο γνωμοδότηση και η συγκήτρια δεν μπορούσε να τις περιλάβει όλα εξ αρχή. Προσωπικά, εγώ θα είχα κάποια πρόταση να υποβάλω, αλλά στα αγγλικά για την απλούστευση. Λαρά θα πήγαινα λίγο πιο μακριά, καθώ οι περισσότεροι συμμετέχοντε που συμμετέχουν σε αυτά τα project ε, παραπονιούνται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο διοικητικό άχθο ε, που οδηγεί σε ε, πολύ λίγη έρευνα. Αν θέλουμε οι μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει να συμπεριληφθούν καλύτερα σε τέτοια project, καινοτομία και έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πραγματικοί εταίροι για να διευκολύνουμε κολλήνουμε τη διάδοση των αποτελεσμάτων και την απλούστευση ε, στην αγορά. Θα πρέπει να είναι αυτή η λέξη κλειδιά, δηλαδή θα πρέπει εκεί ε, να συμμετέχουν όλοι οι ακαδημαϊκοί και οι επιχειρηματίες και ερευνητέ έχουν καλύτερα πράγματα να κάνουν από το να συμπληρώνουν χαρτιά. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να μειώσουμε το άχθος ε, της υποβολής εκθέσεων. Εγώ θεωρώ ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι να διασφαλίσουμε την κατάλληλη διαχείριση αυτών των κονδυλίων, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ του ελέγχου των δαπανών και τι ανάγκης των ερευνητών και των επιχειρηματιών. Η δεύτερη ιδέα που θα ήθελα να δώσω στην γνωμοδότηση θα ήταν μια αναφορά στι προεμπορικέ δημόσιε συμβάσει. Κάτι τέτοιο είναι κάπως επικίνδυνο γιατί κανεί δεν ξέρει αν τελικά το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρχει μια βιώσιμη εφαρμογή στην αγορά και αν θα οδηγήσει σε επένδυση. Έτσι λοιπόν γι' αυτό αυτέ οι προεμπορικέ δημόσιε συμβάσει μπορεί να είναι μια λύση να υπάρχει επιμερισμό του άχθου μεταξύ επιχειρήσει και δημοσίων αρχών. Επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών. Και τέλο, ε, η έκθεση για την νέα αγορά για τι επιχειρήσει και την ανάπτυξη που εθετήθηκε για την δική μα επιτροπή κάλεσε την Κομισιόν να διερευνήσει τη δυνατότητα να συστήσει ένα ειδικό ταμείο επιχειρηματικού κεφαλαίου ε, για ε, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και για ένα πρώιμο στάδιο επενδύσεων. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε αυτή τη γνωμοδότηση. Σα ευχαριστώ και συγχαρητήρια και πάλι για το σχέδιο γνωμοθέτησή σας. Ευχαριστώ, κυρία Ρούλε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Εξαιρετική βάση και περιέχει πολύ καλές νέες ιδέες και εξήγησε πως ε, ε, δεν έχει αρκετό χρόνο για να, χώρο για να επεκταθεί σε αυτά τα οποία θα ήθελε να πει πράγματι αλλά νομίζω καλό είναι να αναφέρει ορισμένα θέματα π.χ. το πώς θα συμπεριληφθεί πραγματί εντονότερα να συμπεριληφθούν εντονότερα και οι δημοσιοπρομηθείες όχι μόνο οι προεμπορικές αλλά και η δυνατότητα εναλλακτικών πρόσφορων Υπάρχουν ε, διάφορες μέθοδοι. Γενικά νομίζω πως θα πρέπει να απλοποιηθούν οι προμηθειες οχι μονο οι προεμπορικες αλλα και η δυνατοτητα εναλλακτικων προσφορων υπαρχουν προμήθειες και να μειωθεί η διοικητική πίεση για να έχουν και οι δύο πλευρές ε, χώρο ελεγμών. Και χαιρετίζω αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Μπουζόη για το διοικητικό βάρος. Ξέρετε και στα διαρθρωτικά ταμεία, σε όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία, υπάρχει μεγάλος σκόπος για μικρά έργα. Και εκεί πέρα μπορεί ίσως να μειωθεί. Κάτι το οποίο θα ήθελα να αναφέρω η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτό το να διαλέγουμε ό,τι μας αρέσει, ε, είναι κάτι το οποίο προκύπτει συνεχώς. Πρέπει να βρεθεί νομίζω μια καλύτερη μέθοδος για να το εμποδίσουμε, γιατί σε πάρα πολλές από τις απαντήσεις στην πράσινη βίβλο αναφέρεται πως αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Τελευταίο. Καλό είναι από το Κοινοβούλιο να λέμε πως θέμε πρωτοβουλίες για συμβάσεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, αλλά αν δείτε τα πραγματικά νούμερα, διαπιστώνουμε πως ε, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα φανταζόμαστε. Αντιθέτως, ειδικά στον καιρό της κρίσης έχουν μειωθεί. Και αυτό σχετίζεται με το κατανομή του κινδύνου νομίζω, που δεν είναι τόσο ξεκάθαρη στη συμπράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και άρα χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο αυτό το μέσο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια. Εγώ θα μιλήσω στο τέλος του πρώτου γύρου, ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η ικανότητα της να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για να αντικαταστήσει όσες χάθηκαν στην κρίση, έγκυται στην ικανότητα της να προωθήσει την καινοτομία στα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και τις κοινωνικές διαδικασίες και πρότυπα. Γι' αυτό και η στόχευση μας θα πρέπει να είναι προς την διευκόλυνση των διαδικασιών χρηματοδότησης, ώστε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υπερβούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία ανάληψης χρηματοδότησης και ταυτόχρονα να βρούμε τρόπους ενθάρρυνσης της χρήσης καινοτόμων λύσεων. Επικεντρώνομαι στις μικρομεσαίες γιατί πέραν το ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση και είναι κατά κανόνα πιο δύσκολη η άντληση επαρκών πόρων. Πέραν από τα όσα έχει προτείνει η συγγήτρια, την οποία και ευχαριστώ για τις πάρα πολύ καλές βασικές της προτάσεις, θα πρέπει να ενσκύψουμε και στην καλύτερη διάρθρωση μεταξύ τοπικών και περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας, με σεβασμό προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων περιεχομένων και ταυτόχρονα ε, και να ενισχύσουμε τις δυνατότητες συντροματικότητας και συνεργασίας μεταξύ τους. Επιπροσθέτως, η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις προεμπορικές συμβάσεις οι οποίες επιλύουν ζητήματα που αδυνατεί να καλύψει η αγορά ή οι λύσεις που προτείνονται είναι ασύμφορες. Ιδιαίτερα για την αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα και την εισαγωγή προσβάσιμων και ευκολόχρηστων υπηρεσιών που παρέχει το κράτος στους πολίτες, είναι αναγκαία η χρήση τεχνολογικά αναβαθμισμένων προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένων για αυτές τις χρήσεις. Καμιά κοινή στρατηγική δεν μπορεί να επιτύχει αν οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν συνεχώς οποιαδήποτε και αν είναι η στρατηγική για την αντιμετώπιση της σημερινής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, οι επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία δεν θα μπορούν να εξασφαλιστούν όσο θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν ανισότητες και ανισορροπίες στην πρόσβαση στα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Ξανά ευχαριστώ την εισηγήτρια και θα επανέλθουμε με τροπολογίες εν ευθέτω χρόνο. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Τριαντεφυλλίδη. Να κάνω και εγώ κάποια σχόλια γιατί ο Σλιφ Φόξ ο εισηγητής δεν μπόρεσε να έρθει. Οπότε να πω και κάποιες παρατηρήσεις ε, της κυρίας Κρεμιά και κάποια δικά μου. Η κυρία Κρεμιά νομίζω έχει επιτύχει εδώ πέρα μια σωστή ισορροπία για την κρίσιμη σημασία αυτής της διαβούλευσης για την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας γιατί γνωρίζουμε πως ε, πρέπει να έχουμε μια πιο καινοτόμο οικονομία και επίσης πως η ευρωπαϊκή έρευνα είναι πολύ υψηλής ποιότητας αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να μεταφραστούν αυτές οι ιδέες σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και να αναπτύξουμε τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για να γίνει αυτό. Και νομίζω πως η ιδέα αυτή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και ε, καλωσορίζω ιδιαίτερα το ότι η Κομισιόν εδώ πέρα κοιτάει ευρύτερα τα πράγματα και κοιτάει ας και τα περιφερειακά κονδύλια και τα κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης γιατί πάρα πολλές ε, καινοτομίες πρέπει να πάνε και στις, ε, στην οικονομία της υπαίθρου. Νομίζω λοιπόν πως ένα από τα πιο σημαντικά Αυτά είναι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά έγγραφα που αφορούν τη στρατηγική 2020 παρά τον έτσι, βαρετό τίτλο που δεν ανταποκρίνεται στη σημασία του πράγματος. Οπότε το καλωσορίζουμε και καλωσορίζω το ότι η Κομισιόν δικαίως ε, άσκησε επικοδομητική κριτική για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της ε, προσέγγισης αυτής και ιδιαίτερα καλωσορίζω και νομίζω πρέπει αυτό να το ενσωματώσουμε σε κάποιες τροπολογίες στην εκθέση Κρέμη, πως η στρατηγική μας είναι ε, να συμβάσουμε την ιδέα των καλύτερων εταιρικών σχέσεων μεταξύ ερευνητών και πανεπιστημίων και εταιριών που έχουν επίσης ιδέες ε, να συνεισφέρουν σε αυτή τη διαδικασία και πιθανούς εταίρους εκμετάλλευσης αυτής της έρευνας και όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και ιδιαίτερα ως πελάτες. Και εδώ πέρα βεβαίως δεν θα σας προξενήσει εντύπωση αυτό δεδομένη συνεργασία μου με την κυρία Ρούλιο και Μπουζόη πως χρειάζεται πράγματι η εμπλοκή των δημοσίων προμηθειών για να βρεθούν πελάτες για αυτές τις τεχνολογίες οι οποίες θα ανταποκριθούν σε ανάγκες της κοινωνίας. Οπότε Νομίζω πως αυτή η ιδέα ενθάρρυνσης των ιδεών και όπως λέει εδώ πέρα να δώσουμε την απαραίτητη ευελιξία και για δημιουργικότητα και διεπιστημονική έρευνα είναι οπωσδήποτε κρίσιμη και θα πρέπει νομίζω βέβαια να ευθυγραμμιστούν ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές αλλά είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση, όπου οι εθνικές κυβερνήσεις και ερευνητές έχουν ε, φοβερές ιδέες, αυτές μπορούν να μεταφερθούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχει κανείς μονοπόλιο στις ιδέες και πρέπει να δούμε και την ποιότητα των ιδεών και το πώς θα μπορέσουμε να τις εκμεταλλευτούμε. Για τις κρατικές ενισχύσεις, νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό αυτό, μόλις πως ήδη η Κομισιόν εξετάζει το θέμα αυτό, οπότε θα πρέπει ε, να μην μας διαφύγει αυτό και όσον αφορά τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων ε, ομάδων καλό είναι να μην περιγράφουμε πάρα πολλά τα πράγματα. Αν υπάρχει ένα γενικό περιβάλλον εντός το οποίο ενθαρρύνουμε τον δυναμισμό θα έρθουν και νέες ομάδες ανθρώπων και εταιρείε νέες και ιδιαίτερα το να προσπαθούμε να βρούμε ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να εμπλακούν και το να αντιμετωπίζουμε κάποια από τα διοικητικά εμπόδια και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες εταιρείες νομίζω αποτελούν συστατικό μέρος αυτής της διαδικασίας. Οι δε σε αυτές και κοινέ τεχνολογικές πλατφόρμες όπου συνεργάζονται οι άνθρωποι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεργάζονται με μεγάλες εταιρείες και μπορούν να τους πουλήσουν ιδέες είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Είμαι ικανοποιημένο για την αναφορά που έγινε στην πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλω να πω κάτι γρήγορα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Είναι σαφές πως ε, το Ευρωπαϊκό αυτό Ινστιτούτο που είχε στόχο αυτό το οποίο πρότεινε η κυρία Γκίγεν Κουίν πρέπει νομίζω να ενσωματωθεί σε ολόκληρη αυτή την Ένωση καινοτομία. Και μου φαίνεται πω θα ήταν πάρα πολύ λογικό να υπαχθεί στη Γενική Διεύθυνση έρευνα γιατί εκεί πέρα νομίζω θα συνεισφέρει τα μέγιστα. Και θα πρέπει να είμαστε σαφείς για την ε, εντολή του. Μέρος της εντολή του είναι να ερευνήσει και να αναπτύξει μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίες και εμείς θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ε, συμμετέχοντες ε, στις κοινότητες της γνώσης και της καινοτομίας να πειραματίζονται με νέες ιδέες για τη μεταφορά της τεχνολογίας. Κατά την άποψή μου πρόκειται περί ενός εργαστηρίου ανάπτυξης των διαδικασιών αυτών, να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε τις δημόσιες προμήθειες, να δούμε πώς θα βρούμε τα οργανωτικά εκείνα παραδείγματα για κοινέ τεχνολογικές πλατφόρμες και ελπίζω στη νέα στρατηγική του Ινστιτούτου αυτού να δούμε αυτό το ενδιαφέρον γιατί αυτό κατά την άποψή μου θα πρέπει να αποτελεί κύριο στόχο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και θα καταθέσουμε και κάποιες τροπολογίες σχετικά. Οπότε θεωρώ πως ε, είναι μια συναρπαστική ευκαιρία αυτή για την Επιτροπή μας ε, να βάλει εδώ τη φραγίδα της και για να ολοκληρώσω ένα από τα θέματα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η αμοιβή αναγνώριση προσόντων. Η Κομισιόν εδώ πέρα μας ε, ρωτάει για πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν στην κοινή ευρωπαϊκή, στον κοινό ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο. Και η κυρία Γκίγκεν Κουίν λέει πως υπάρχουν εμπόδια στην αμοιβαία αναγνώριση, στην απασχόληση που εμποδίζουν τους ερευνητέ να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο. Αυτό πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε και να συνεισφέρουμε εδώ πέρα και την δική μας βοήθεια. Και οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, ε, το οποίο ήταν μεγάλη επιτυχία, ήταν επιτυχημένο γιατί εστίασε αποκλειστικά στην ποιότητα των συνεισφορών μεμονωμένων ερευνητών. Γνωρίζω πως κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή κάποιες ιδέες για να μειωθεί να μειωθούν οι αρμοδιότητες του. Εγώ θεωρώ πως πρέπει να επιμείνουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας ε, ως ε, μια διαδικασία με κινητήριο δύναμη την ποιότητα όπου υποστηρίζονται οι πιο ποιοτικέ έρευνες γιατί αυτή η έρευνα νομίζω θα κινητοποιήσει την όλη διαδικασία καινοτομία. Τώρα από τους υπόλοιπους ομιλητές κυρία Βανιού, κάποιος άλλος Μπερνατέτ ευχαρίστως να σας δώσω τον λόγο Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη γιατί ακούσαμε ήδη πάρα πολλά πράγματα και δεν θέλω να τα επαναλάβω. Θα ήθελα να συγχαρώ τη Λάρα για την εξαιρετική δουλειά που έκανε και πόσο μιλούσε για νέους και για γυναίκες. Θεωρώ ότι η ικανότητα καινοτομία που έχει και ο ενθουσιασμό που τη διακρίνει αντισταθμίζει αυτή την απογοήτευση βαθιά που ένιωθε διότι δεν μπορούσε να συντάξει ένα ογκώδε κείμενο όπω θα ήθελε. Πάντως, για την έρευνα η αρχή της έκθεσης ήδη είναι εξαιρετική βλέπουμε ότι επιτόπολα συμβαίνουν σε επίπεδο περιφερειών. Οι περιφέρειες καινοτομούν με τα ιδρυτικά ερευνητικά τους κέντρα, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι τα φυτόρια της συνεργασίας και της καινοτομίας. Ε, άρα έχει θεμελιώδη σημασία αυτό το ζήτημα. Μέσα από τα ερευνητικά προγράμματα να προωθήσουμε τη συνεργασία και κατόπιν να τα συνδέσουμε με τα ταμεία συνοχής. Εάν υπάρξει κατάλληλη συνεργασία, θα υπάρξει και ορθή χρήση των κονδυλίων, των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχή και θα ενισχυθεί η συνοχή στο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θα ήθελα να σχολιάσω αυτέ τι ε, συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Θα συμφωνήσω βέβαια με τα σχετικά στοιχεία τη έκθεση, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η έννοια τη συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα λόγω τη κρίσης ε, και κατόπιν χρειαζόμαστε επιμερισμό κινδύνων, ναι μεν, αλλά ουσιαστικά πολλαπλασιάζουμε τις ε, σχέσεις αυτές ε, και δεν τις καθιστούμε πιο πιο ποιοτικέ απαραίτητα. Χρειάζεται επίση νομική ασφάλεια που να πλαισιώνει αυτέ τι σχέσει, ώστε να διεξάγονται προ όφελο ε, των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και των κρατών τη Ένωση. Κάτι άλλο που από ό,τι κατάλαβα δεν συμπεριλάβατε στην έκθεση ε, λόγω περιορισμού είναι το θέμα του διπλώματο τεχνία, του ευρωπαϊκού διπλώματο ευρεσιτεχνία. Είναι μία ξεκάθαρη έννοια. Υπάρχει κατοχήρωση αλλά όχι επαρκής προς το παρόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να ενισχυθεί αν θέλουμε ε, να ενισχυθούν οι περιφέρειες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα επωνομαζόμενα κλάστερς, οι ομάδες, ε, έχει λειτουργήσει σωστά ε, η ιδέα αυτή. Το ίδιο και οι Watchers. Νομίζω πρέπει, μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή την ιδέα όπως μας είπε και ο Μάλκολμ κυρίως σε επίπεδο κινητικότητας των ερευνητών ε, ε, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που μας χρειάζεται είναι μια ξεκάθαρη άποψη, μια συνενετική άποψη ως προς τα επαγγελματικά προσόντα. Όταν διασχίζει κάποιος τα σύνορα και πάει να εργαστεί σε ένα άλλο εργαστήριο, τι χρειάζεται, τι απαιτείται. Να είμαστε ξεκάθαροι ούτω ώστε στον τομέα της ε, καινοτομία να έχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Μπορώ να μακρηγορίζω, δεν έχουμε χρόνο. Εξαιρετική δουλειά έκανες Λάρα και σε συγχαίρω και πάλι κλείνοντα. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κρότσμαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την Λάρα ακόμη, γιατί έδωσε βάρος μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν προϋπολογισμό έρευνας, δεν έχουν πρόβλημα να κάνουν έρευνα και να την εφαρμόσουν κιόλας. Ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δυσκολία να βρουν ερευνητικά κονδύλια και αν θέλουν να λάβουν τέτοια κονδύλια υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία και δεν έχουν άρα την εμπειρία και βεβαίως έχουν πάντα προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή αυτής της έρευνας στην παραγωγή έτσι να καταταλήξουν σε ένα προϊόν. Ξέρουμε λοιπόν πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνες οι οποίες ε, είναι αν θέλετε τα, τα χύπλοα που θα κινηθούν πιο γρήγορα και όχι μεγάλες που θα χρειαστούν χρόνο για να εφαρμόσουν κάτι. Και νομίζω πως αυτό μετά θα δώσει και μια όθηση στην ε, εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ να δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Κρός για να σχολιάσει. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά να ακούσουμε και δική σας άποψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα και άκουσα αυτή την πολύ επικοδομητική συζήτηση για όσα σωστά είπατε θα είναι μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση για ένα σημαντικότατο θέμα. Νομίζω ότι ορθά ε, είπατε ότι το κοινό στρατηγικό πλαίσιο σκοπεύει να ομαδοποιήσει μια σειρά δραστηριοτήτων υπό μια κοινή ομπρέλα και πραγματικά εμείς επιζητούμε να θέσουμε τον αντίκτυπο των δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ταυτόχρονα να υποβάλουμε σε ένα νέο πλαίσιο όλα αυτά, πλουστεύοντας τους κανόνες και δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που θα είναι πιο φιλικό προς το χρήστη. Άκουσα τα σχόλιά σας, πολλοί από εσά και η κυρία Κόμη αναφέρθηκε στη σημασία του συνδεσμού με την πολιτική συνοχής και συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να προσδιορίσουμε συνέργειες με τα διαρθρωτικά ταμεία. Θέλουμε όμως να πούμε ότι εδώ μιλάμε για ξεχωριστές πολιτικές και εμείς ε, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα καινοτομία και έρευνά έχει ως κατευθυντήρια ε, δύναμη το θέμα της αριστείας. Όμως ε, παρόλα αυτά όλα τα μέρη της Ένωσης θα βρίσκουν το χώρο τους και τη θέση τους στο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Αναφερθήκατε και σε κάποια άλλα ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη το να χρησιμοποιούνται κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Ε, αυτά είναι θέματα τα οποία τα εξετάζουμε και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και αφορούν τομεί ε, που φυσικά θα διερευνήσουμε και θα δούμε σε ποιο βαθμό μπορούν να συμπεριληφθούν αυτά στο πρόγραμμα. Όπως γνωρίζετε, η Πράσινη Βίβλος, ε, με την Πράσινη Βίβλο ξεκίνησε μια μεγάλη διαβούλευση, η οποία έχει τώρα ολοκληρωθεί, αλλά να σας πω ότι είχαμε 1.300 απαντήσεις στο επιγραμμικό ρητοματολόγιο και είχαμε και 700 έγγραφα θέσεις που κατατέθηκαν από τους διάφορους συμμετέχοντες, από τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και υπήρχε και ένα σκεπτικό στρατηγικής που το βρήκαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θεωρούμε ότι τώρα αυτή η πολιτική είναι όρημη και πραγματικά το τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από όλη την Ένωση μας έδειξε τι αντίκτυπο μπορεί να έχουμε με αυτό το νέο πρόγραμμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης υπάρχει στην Ένωση όχι μόνο να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο για όλες αυτές τις δράσεις αλλά και για τα θέματα που θέσατε σήμερα το απόγευμα και φυσικά για την ανάγκη απλούστευσης. Εμείς ε, την Παρασκευή ολοκληρώσαμε τι διαβουλεύσει με ένα μεγαλύτερο εδώ στις Βρυξέλλες ε, τώρα συστήνουμε, εκπονούμε τις προτάσεις μας για το νέο πρόγραμμα. Το πλήρες πακέτο θα κατατεθεί μέχρι τα τέλη του έτους, οι πλήρες δέσμοι μέτρων. Και για το όνομα, σωστά το είπατε, είναι κάπως διοικητικό. Έτσι λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε τώρα ένα διαγωνισμό. Ε, υλοποιούμε ένα διαγωνισμό για να έχουμε ίσως ένα νόημα, ένα όνομα που να σημαίνει περισσότερα και θα καταλήξουμε και σε ένα κατάλογο για πιο φιλικές ονομασίες του νέου προγράμματος. Σας ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Χαίρομαι πάρα πολύ που οι ιδέες μας για τις προκλήσεις ε, συμπεριλαμβάνονται και στο δικό σας σκεπτικό. Χαίρομαι πάρα πολύ επίσης που οι φίλοι μας από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ιστορικής Αγοράς και από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Enterprise ε, συμμετέχουν. Λοιπόν, να ξαναδώσουμε το λόγο στην κυρία Κόμη για να συνοψίσει και να επιβεβαιώσει και το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τις συνεισφορές σας και σήμερα αλλά και τις προηγούμενες ημέρες Ευχαρίστησα και τον κύριο Μπουζόη για το ότι είναι τόσο ανοιχτό και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ που παρενέβηκε στα Ιταλικά. Ε, ο στόχος είναι να έχουμε μια έρευνα που θα προσανατολίζεται στην αγορά, δηλαδή μια έρευνα που να είναι πραγματικά λειτουργική για τον πολίτη και να μην βασίζεται στα μέγιστα συστήματα που κατόπιν στην καθημερινή ζωή δεν χρησιμοποιούνται και πάρα πολύ ή θα χρησιμεύσουν ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι ο στόχος. Το η άλλη για την απλούστηση Βλέπω ότι πολλοί από εσά ε, εξάφρασαν κάποιες ανησυχίες για το θέμα αυτό. Εγώ έρχομαι από μια χώρα όπου η απλούστευση είναι πάντοτε στην ημερησία διάταξη γιατί υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία στη χώρα μου. Έτσι λοιπόν, αν τελικά ε, κατορθώσουμε να έχουμε κάτι τέτοιο ε, σε ένα περιφερειακό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει απλούστευση γιατί είμαστε πιο κοντά στο πολίτη και πιο κοντά στις επιχειρήσεις. Αυτή η ιδέα να μεταβούμε από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο, στο περιφερειακό επίπεδο, γιατί και για τα βάτσερ και τα κουπόνια αυτά υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια γιατί ο έλεγχο γίνεται είτε από τι περιφέρειες είτε από την Επιτροπή. Γιατί ε, είναι διαπιστευμένα τα ερευνητικά κέντρα αλλά γίνεται και αξιολόγηση από την ίδια την αγορά. Γιατί ε, αν λειτουργεί αυτή η έρευνα τότε γίνεται ίδια δοκιμή από την αγορά. Βλέπουμε αν είναι προσανατολισμένη η έρευνα στην αγορά. Εγώ μπορώ να σα πω ότι εξεπλάγει είναι ευχάριστα από την ενότητα με την οποία εκφράστηκε η Επιτροπή ΙΜΚΟ σήμερα, αλλά και για τι προτάσει που κατατέθηκαν. Έτσι λοιπόν, ε, να καταθέσω εδώ μία μικρή πρόκληση, γιατί είμαι και μέλο τη Επιτροπή Βιομηχανία. Μία σκέψη ε, στο να υπάρχει και μία μεγαλύτερη συνεισφορά ε, τη Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά. Αυτό βέβαια θα το δείτε εσεί. Εγώ σα προκαλώ γιατί όπως βλέπετε ε, ίσως τώρα είναι πιο επικοδομητικό το κλίμα από ό,τι άλλες φορές. Εμείς ε, φυσικά θα συνεισφέρουμε τα μάλλα γιατί πιστεύουμε σε μια ευρωπαϊκή έρευνα, σε μια έρευνα που να ενισχύει την ενιαία αγορά. Εγώ επιβεβαιώνω όλες τις ημερομηνίε που είχαμε καθορίσει, δηλαδή προθεσμία για τις τροπολογίες ε, 22 Ιουνίου την επόμενη εβδομάδα και εγώ είμαι φυσικά στη διάθεσή σας 22 λέει ο μιλήτρια 21 21, 21 Ιουνίου να έχουμε μία ενότητα της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και με τις τροπολογίες. Νομίζω αν είμαστε ενωμένοι αυτό θα βαρύνει πολύ διαφορετικά στην Επιτροπή Βιομηχανίας και θα έχει και διαφορετική αξία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πράγματι 21 Ιουνίου 12 το μεσημέρι. Και θα συζητήσουμε τις τροπολογίες 12 Ιουλίου και θα ψηφίσουμε 12 Ιουλίου και μετά θα πρέπει βεβαίω να πείστε και την Επιτροπή Βιομηχανίας γιατί αυτοί θα ψηφίσουν 30 Αυγούστου. Αλλά συμφωνώ πως είναι σημαντικό. Έπρεπε να το είχα πει και πριν. Καλωσορίζω και τον κύριο Σίπεν, την κυρία Σίπεντς από την Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας των Πληροφοριών και είχαμε συνεργαστεί βεβαίως και για την προεμπορική τις προεμπορικές δημοσιοπρομηθίες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και περνάμε στον προϋπολογισμό και Χαίρομαι που καλωσορίζω τον Έντβαρτ Κόσνικη, συγητή μας για τον προπολογισμό και βεβαίως έχουμε κάποιους ε, σκιοδησηγητές. Βλέπω τον κύριο Ντεκάμπους εδώ πέρα για το ΕΛΚ. Δεν ξέρω η κυρία Γκέπχαρτ ε, ε, ποιος θα παρακολουθήσει τον προπολογισμό για τους σοσιαλδημοκράτες. Κυρία Γκέπχαρτ, μας ακούτε. Κάποιος από τους σοσιαλδημοκράτες θα παρακολουθήσει τον προπολογισμό. Ο κύριος Μπουζόη, α, ο κύριος Κρόιτσμαν. Κυρία Ρούλε, θα πει κάτι για τους πράσινους και ο κύριος Τριανταφυλλίδης είναι εδώ. Λοιπόν, κύριε Κοσίσνικ, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, πριν περάσω στην ουσία του ζητήματος που μας απασχολεί, Εξάλλου όλοι έχετε εμπλακεί σε μικρότερο σε μεγαλύτερο βαθμό σε αυτή την υπόθεση. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τις τελευταίες εξελίξεις για την έγκριση του προϋπολογισμού. Κύριος Γαμποσάνη, συγγετής για το σχέδιο προϋπολογισμού, ηγείται όλων των προσπαθειών που γίνονται και τώρα ήρθε η στιγμή να ε, συντάξουμε τη δική μας γνωμοδότηση. Ε, συναντήθηκα με τη Φραντζέσκα Ποζόνη και τον κύριο Λαμασού σήμερα το πρωί. και συναντηθήκαμε εξάλλου και με τους λοιπούς εισηγητές των υπολείπων δηλαδή επιτροπών για μια ανταλλαγή απόψεων και θα ήθελα να συνοψίσω το περιεχόμενο των συζητήσεών μας. Συζητήσαμε τα περί ε, τριμερούς διαλόγου που έχει προγραμματιστεί για την 11η Ιουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ημερομηνία αυτή για μας. Ο κύριος Λαμασούρ και ο εισηγητής είπαν ότι αν ναι, οι μεμονωμένες επιτροπές παρουσιάσουν πιλωτικά προγράμματα και θελήσουν να προωθήσουν τα δικά τους πιλωτικά προγράμματα. Γίνεται δεκτό αυτό ε, και οι υπόλοιπε επιτροπές μπορούν να υποβάλουν σχετικές τροπολογίες μέχρι την 11η Ιουλίου. Ας περάσω τώρα στην γνωμοδότησή της Επιτροπής μας. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων ε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και φαίνεται ότι καταλήξαμε σε κάποια συμφωνία σχετικά με τις ανάγκες μας. Η μεγαλύτερη ανάγκη που έχουμε είναι μια εξορθολογισμένη προσέγγιση, ούτω ώστε να απορροφούνται με τον πλέον ε, αποτελεσματικό τρόπο όλα τα κονδύλια και να βελτιωθεί έτσι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Υποστηρίζουμε την πράξη για την ενιαία αγορά, θεωρούμε ότι θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα, όλα αυτά τα αναφέρω μέσα στην έκθεση. και συμφωνούμε με την τοποθέτηση του Επιτρόπου Μπαρνιέ για αυτό το θέμα. Επίσης, Υποστηρίζουμε και την ιδέα του φόρουμ της ενίας αγοράς μέσα στη γνωμοδότηση. Σίγουρα θα συμφωνήσετε ε, και εσείς μαζί μου γιατί εσείς είχατε την ιδέα. Είναι σαφές ε, ότι δεν θα χρηματοδοτηθούν ε, όλα τα προγράμματα όπως τα θέλαμε και ε, αναφερόμαστε στις περικοπές δαπανών που έχουν γίνει στο πρόγραμμα Solvit. Ε, θα δείτε τις λεπτομέρειες στους φακέλους σας. Ε, θέλω όμως να σχολιάσω τώρα την 20η Ιουλίου που είναι η ημερομηνία, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών για αυτά τα νέα σε εισαγωγικά προγράμματα. θα πρέπει όλοι να λάβουμε υπόψη τη, το κλίμα που επικρατεί στον προϋπολογισμό λόγω κρίση, ε, πριν το αποθετηθούμε, πριν υποβάλουμε τροπολογίες. Θα ήθελα τώρα να ακούσω τις δικές σας απόψεις για να συμπεριλα... τι συμπεριλάβω στη γνωμοδότηση. σας. ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος. Ήσασταν σαφέστατος και είναι σαφή και η έκθεσή σα. Έχουμε και συγκεκριμένα με μονομένα σημεία που μας καλείται να εξετάσουμε. Θα περάσουμε σε αυτό. Ας δούμε τους σκιώδες εισηγητές πρώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω πέντε σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, ευχαριστώ τον εισηγητή του για τις ξεκάθαρες ε, συμβουλές του. Νομίζω πως είναι σαφές ποια είναι η διάθεση εδώ της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και έρχομαι άρα στη δεύτερη παρατήρησή μου. Την προηγούμενη εβδομάδα παρατήρησα πως ε, ε, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό ε, προϋπολογισμό για το αν χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και αν ε, πρέπει να αυξηθεί κτλ. Και, πράγματι αυτό ελήφθη υπόψη τρίτον. Η παρατήρηση επί του σημείου 3, ε, Single Market Act, 12 ε, μοχλή για να ανάπτυξη και εμπιστοσύνη. Ο εισηγητής θεωρεί πως ο προϋπολογισμός επαρκεί για κάτι τέτοιο. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Ωραίο είναι ε, που παρουσίασε ένα τέτοιο σχέδιο ο Επίτροπος Μπαρνιά, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά. Με τις ε, προθέσεις ε, δεν κάνουμε τίποτα και το ερώτημα είναι κατά πόσον έχει μετρήσει κάτι τέτοιο, γιατί μιλάει μόνο για μία μικρή αύξηση για την εφαρμογή του προγράμματος. Επαρκεί αυτό. Κατόπιν, για το φόρουμ της ενιαίας αγοράς, ε, ξέρετε πως εντωμεταξύ έχουμε δύο προκαταρκτικές προτάσεις που έχουμε λάβει. Συμφωνώ πως ε, το φόρουμ ε, της ενιαίας αγοράς ε, που θα λάβει η χώρα στην Κρακοβία πρέπει να το στηρίξουμε και θα κατατεθεί σχετική τροπολογία ταυτόχρονα και αυτή είναι η πέμπτη μου παρατήρηση είναι κρίμα να κάνουμε οικονομίες στο Solvit και το ερώτημά μου απευθύνεται προς τον εισηγητή αλλά οπωσδήποτε και τους συναδέλφους Κρόιτσμαν και Σχαλτεμόζετ το εάν το πιλωτικό αυτό έργο, τα, έργα, τα λεφτά του πιλωτικού έργου μπορούν να πάνε στο Solvit. Δεν ξέρω, μπορεί να μην συμφωνεί με τους κανόνες του προπολογισμού. Αλλά γιατί ξεκινάμε καινούρια πιλωτικά έργα τη στιγμή που κόβουμε από το Solvit. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φαντεκάμπ. Κρόιτσμαν και να δούμε αν θα μιλήσει για από τους σοσιαλδημοκράτες. Α, κυρία Σχαλεμόζα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κουσούσνικ για το σχέδιο έκθεσης που αντιμετωπίζει τα πιο σημαντικά ζητήματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας. Καλώ ορίζουμε την προσέγγιση του εισηγητή όταν λέει πω ο προπολογισμό της Ένωσης πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία τη οικονομική ανάπτυξη και για τον σκοπό αυτό τα κονδύλια πρέπει να πάνε στους τομείς εκείνους και τις επενδύσεις που συνεισφέρουν στην οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Επίσης πρέπει να έχουμε κατά νου πως ζητάμε και τις εκθέσεις της πράξης της εσωτερικής αγοράς και τις 12 μοχλούς αυτούς της Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν οι τίτλοι 1 και 3 να αντικατοπτρίζουν αυτές τις ε, προτεραιότητες. Επίσης ανισχούμε για την μη κατανομή των κονδυλίων για το Solvit, καθώς το Solvit αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην Ένωση. Επιπλέον η αξιολόγηση που έχει γίνει μέχρι στιγμή αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα και την προσθέμενη αξία του, άρα αποτελεσματικά ξοδεύονται τα λεφτά σε αυτόν τον τομέα. Γι' αυτό η Επιτροπή μας πρέπει να παλέψει για επαρκείς πόρους για το Solvit και τις λοιπές υπηρεσίες της εσωτερικής αγοράς για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να βοηθούν τους πολίτες μας. Οπότε στηρίζει τις προτάσεις ε, του εισηγητή για να πάνε λεφτά σε αυτή τη γραμμή του προπολογισμού. Το ίδιο ισχύει και για το φόρουμ το, της κοινή αγοράς, το πιλωτικό αυτό έργο. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν και την Πολωνική Προεδρία για την διοργάνωση ε, του φετινού φόρουμ. Βεβαίω δεν μπορούμε να προβλέψουμε την επιτυχία τη εκδήλωση, αλλά ο κ. Μπουσόη είναι πεπισμένο πω το φόρουμ εσωτερική αγορά θα χρησιμεύσει για να τονίσει τι μεγάλε ανησυχίε των πολιτών μα και επιχειρήσεων και να τι θέσει στο πολιτικό προσκήνιο. Έτσι έχουμε μια ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά οι πολίτες και επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά και άρα πρέπει να επιμείνουμε στην χρηματοδότηση του φόρουμ της εσωτερικής αγοράς της ενιαίας αγοράς για το οποίο δεν έχει προτείνει τίποτα η Κομισιόν και θα ήθελα να προσθέσω κύριε Κοσουσνίκ πως ε, προτείνετε εσείς και η κυρία Σχάλντεμος ε, μία τροπολογία για ένα έργο για τις αρχές επιτήρησης αγοράς. Είναι σημαντικό αυτό. Κάθε φορά βλέπουμε πως ε, κάνουμε προτάσεις και δεν υπάρχει αρκετή επιτήρηση της αγοράς. Και αν δεν έχουμε καλύτερες ε, λύσεις για την επιτήρηση της αγοράς φοβούμε πως όλες οι τροπολογίες, όλοι οι κανονισμοί που περνάμε εδώ δεν έχουν ε, νόημα. Γιατί συχνά διαπιστώνουμε πως οι ελλείψεις ε, στην επιτήρηση της αγοράς ε, που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη να ρωτήσει κανείς δηλαδή, διαπιστώνει πως κάποια κράτη-μέλη κάνουν πολύ καλή δουλειά, έχουν αρκετούς ανθρώπους ε, προσωπικό για αυτή τη δουλειά και άλλοι το κάνουν πιο χαλαρά θα έλεγα. Οπότε αυτή είναι η πρόταση που έχουμε καταθέσει από κοινού και χαίρομαι για το ότι την στηρίζετε και πρέπει πράγματι να το προωθήσουμε αυτό. Τόσο δεν θα διαβάσω αυτό το οποίο προτείνουμε, αλλά θα ήθελα να συμφωνήσω και να προσθέσω αυτό στην απόψη του κύριου Μπουσόη. Ευχαριστώ κυρία Σχαλτεμόζε. Man, jeg bliver lige kastet direkte ud i at <laughs> skulle forholde mig til budgettet. Men, øh, men jeg vil først starte med at sige, at det forslag som... Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε η πρόταση την οποία συνυποστήριξα περί πιλωτικών έργων ενίσχυσης της ε, εποπτείας της ε, αγοράς, ε, ξέρετε, δεν είχε στόχο να φύγουν και να κοπούν λεφτά από το Solvit. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε κάποια έμφαση στην εσωτερική αγορά, αλλά αυτό κάτι έξτρα που θα προσθεθεί στα υπάρχοντα, όχι να κόψουμε απαλού. Και είναι κρίμα πράγματι να γίνονται ε, περικοπές στον τομέα της εσωτερικής αγοράς και συμφωνούν όλοι ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη και για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να λειτουργεί εύρυθμα η εσωτερική αγορά. Οπότε πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις ως προς την επιτήρηση της αγοράς. Πρέπει να είμαστε ακόμη πιο σαφείς ε, σε σχέση με αυτό που λέει ο εισηγητής ότι δηλαδή η επιτήρηση πρέπει να αναδειχθεί σε προτεραιότητα. Για να λειτουργήσει, για να επιτύχουμε αυτό το εγχείρημα χρειαζόμαστε σωστή επιτήρηση της αγοράς. Οφείλουμε να τονίσουμε αυτή τη διάσταση. Ε, θα μπορούσαμε ίσως ε, και να προσθέσουμε κάποια στοιχεία, αλλά κατά τα άλλα είναι εξαιρετική η έκθεση. Παρακαλώ λίγα λόγια χαιρετίζω τη νέα πρόταση ανταλλαγών μεταξύ των αρχών εποπτείας αγοράς. Καλή ιδέα και ίσως ο εισηγητής μπορεί να μας εξηγήσει γιατί έχουμε λιγότερα λεφτά για το Solvit. Ε, γιατί δεν εξαντλήθηκαν την προηγούμενη φορά ή απλά περικόπηκαν. Um, Άλλος κανείς, ε, κύριε δεν εκπροσωπείται μάλιστα. Να ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Κοζούνικ να αναφερθεί στα θέματα που ακούστηκαν όπως για το Solvit ε, και να μας πει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ όλους ε, όσους ε, πήραν το λόγο στη συζήτηση. Εγώ θα έκανα μια πιο πολιτική παρατήρηση γιατί τελικά εδώ πολιτικοί είμαστε και νομίζω ότι το δικό μας ενδιαφέρον είναι της διάδοσης και της εμβάθυνσης ε, στην εσωτερική αγορά. Εγώ νομίζω ότι η ενιαία αγορά αποτελεί μία από τις μεγάλες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε πεπισμένοι ότι σε πολιτικό επίπεδο αυτό έχει νόημα για όλους τους πολίτες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης συμφωνώ για το ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου μία σειρά προτεραιοτήτων έτσι ώστε να τις αντικατοπτρίσουμε και σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης, γιατί είναι λογικό ότι η προτεραιότητά μας είναι η νέα αγορά. Και αν θυμόμαστε τι συμβαίνει από την αρχή αυτής της θητείας, όλοι συμφωνούσαμε παρκώς με το ότι τελικά ε, είχε ασκηθεί κάποια κριτική στη σημερινή κατάσταση της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό δημιουργήθηκε και αυτό το φόρουμ για την εσωτερική αγορά, γιατί εκεί επισημαίνονται τα πιο σημαντικά, οι πιο σημαντικές πτυχές. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου μία σειρά και άλλων στοιχείων για τον προπολογισμό όπως τα παράγοντα της Βραζιλίας. Το αυτό το ανέφεραν και συνάδελφοι σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ορισμένοι υποστηρίζουν, παραδείγματο χάρη, την ανάπτυξη για τη Βραζιλία. Και εγώ δεν νομίζω ότι αυτό είναι και το σορθό, γιατί η Βραζιλία δεν είναι μεταξύ των ε, αναπτυσσόμενων χωρών, δεν θεωρείται ω τέτοια. Έτσι λοιπόν υπάρχει μία σειρά παραγόντων που πρέπει να αποσαφηνίσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι με σαφή τρόπο θα πρέπει να θέσουμε τις προτεραιότητες και να τις συζητήσουμε μαζί σας. Σημειώνω όλα τα σχόλια που ακούστηκαν κυρίως ε, σε ό,τι αφορά το Solvit, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω λάβει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η πίεση να μην αυξηθεί ο προπολογισμό για το Solvit, από όσο γνωρίζω, προέρχεται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι από το Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν ε, θα προσπαθήσουμε και εμείς να ασκήσουμε πίεση στην Εκτελεστική Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, μεμονωμένες παρατηρήσεις, δεν ξέρω. Ίσως να αντιδράσω σε κάτι που υπόθηκε από τον συνάδελφο αν θέλουμε, δηλαδή αυτά τα 12, αυτή 12 πόντι, ε, συγγνώμη, αυτά τα 12 σημεία του Επιτρόπου Μπαρνιά θα μας βοηθήσουν στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι εμείς ε, θα πρέπει ε, να λειτουργήσουμε έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει διαφορά εδώ με αυτά τα 12 σημεία. Θα πρέπει να προβούμε και στον κατάλληλο έλεγχο. Σε ό,τι αφορά την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 20 Ιουλίου και φυσικά είμαι ανοιχτό σε οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση για βελτίωση του σχεδίου κειμένου. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να βελτιώνουν τα πράγματα γιατί ε, είναι πολύ καλή επικοινωνία με την κυρία Μπαλτσάνη και εγώ νομίζω ότι είναι ανοιχτή στο να λάβει και τροπολογίε και από τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να τα ξαναπούμε μόνο για το χρονοδιάγραμμα γιατί νομίζω ότι είναι καλό να συζητήσουμε με όλους τους κοιόδης. Ε, προθεσμία για τις τροπολογίες 20 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι, 31 Αυγούστου εξέταση τροπολογιών και ψηφοφορία. Και τότε θα έχουμε και την προθεσμία για την Επιτροπή Προϋπολογισμού 8 Σεπτεμβρίου. Εντάξει. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ε, ευχαριστώ και εσάς, αλλά και τους κοιόδης εισηγητές για το έργο αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πραγματική ευκαιρία να υιοθετήσουμε μια πολιτική προσέγγιση επί τομέων που θα προωθήσουν την ενή αγορά. Τώρα θα περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης, ε, μια παρουσίαση μελέτης που αφορά την τελωνιακή συνεργασία στον τομέα ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, ο ρόλος των τελωνίων στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ζήτησαν αυτή τη μελέτη. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είχαν τα μέλη αυτή τη Επιτροπή ακόμη την ευκαιρία να δουν αυτή τη μελέτη, γιατί είναι πάρα πολύ απασχολημένοι. Αλλά θεωρούμε και εμεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μελέτη και θέλουμε να κατανοήσουμε τι περιλαμβάνεται εκεί, γιατί τα τελωνία είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έτσι λοιπόν, ε, θέλω να καλωσορίσω τον αρμόδιο τη μελέτη αυτή, τον κύριο Κομπίτ, που ήρθε να μα την παρουσιάσει. Δυστυχώς ο κύριος Σαλντίνη που είναι εισηγητής ε, έμεινε στην ε, Ιταλία λόγω του δημοψηφίσματος αλλά είναι εδώ και άλλοι συνάδελφοι όπως Μίθιον που εργάζονται με το φάκελο των τελωνίων εδώ ε, και εγώ ήμουν επίσης και ο για το θέμα αυτό και θα ήθελα να καλωσορίσω και την κυρία Τούρμ ως κοιόδη Ε, η κυρία Κορέλα μου ζήτησε να παρουσιάσω τη δική της θέση, μάλιστα. Είπε η κυρία Τούν. Ε, ναι, θέλω να καλωσορίσω και τον συνάδελφο Σιλένσκι που συμμετέχει στην Επιτροπή μας και είναι αρμόδιος για την τελωνιακή πολιτική και για την ομοθεσία. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ στενά για την έκθεση της κυρίας Σαλντίνη. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Χόμπινγκ είναι ε, ε, μέλος του κέντρου της Ευρωπαϊκής, ε, των μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ε, έχει παράσχει συμβουλές και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Έτσι λοιπόν σας καλωσορίζουμε, έχετε κάποιες διαφάνειες, θα σας δώσω το λόγο για να τις παρουσιάσετε και κατόπιν θα έχουμε ερωτήσεις. Κύριε Χόμπινγκ. Well, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και θέλω να το τονίσω και να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω να σας παρουσιάσω τη μελέτη μου. Προφανώς ε, είναι τιμή για οποιονδήποτε να παρουσιάζει μια έκθεση που συνέταξε σε οποιαδήποτε επιτροπή, αλλά χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που απευθύνομαι ε, σε μια επιτροπή που δεν είναι αυτή που ζήτησε τη μελέτη. Ωραίο είναι, προφανώς ε, δημιουργεί και κάποια προβληματάκια, όπως είδατε από τον τίτλο. Πρόκειται για ε, το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ε, και αυτό δεν εντάσσεται κανονικά στην εντολή της δικής σας επιτροπής, αλλά τι έγινε. Το τελευταίο τρίμηνο σημειώθηκαν αλλαγές και είναι ομιχλώδες το τοπίο όταν ε, μιλάμε για κανονιστικά ζητήματα που αναμειγνύονται. Δηλαδή όταν συζητάτε για θέματα ασφαλείας μπορείτε να δείτε κάποια στοιχεία μέσα στον τον τελωνιακό κανονισμό και το αντίστροφο. Για τα θέματα ασφαλείας προφανέστατα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, στα νομοθετικά κείμενα της Ένωσης. Ε, βρισκόμαστε λοιπόν σε μια νέα φάση ανάπτυξης ε, των νομικών πράξεων για το θέμα των τελωνίων και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ σήμερα. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ελπίζω να μην σας τρομάξω τώρα με αυτές τις διαφάνειες. Ε, ήθελα ως ήθιστε να κάνω μια ιστορική αναδρομή 2.000 ετών. Ε, θα μας πάρει χρόνο από πλευράς δηλαδή ετών, αλλά εγώ θα είμαι πολύ γρήγορος. Ε, θα κάνω μόνο κάποιες ε, στάσεις αλλά θα τα δείτε αυτά στις επόμενες διαφάνειες. Ε, Ελληνορωμαϊκός κόσμος, ε, πάρα πολύ σημαντικό διότι πρώτη φορά τα τελωνία ανέλαβαν τις αρμοδιότητές τους ε, και κλήθησαν να παραγάγουν ιδέες για να εφαρμόσουν το σύστημα που επιθυμούσε, αν θέλετε, η κυβέρνηση. Ε, επίσης, μην ξεχνάτε τι γινόταν με τον Απόστολο Ματθαίο. Ήταν φοροεισπράκτορας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρείται ότι θεωρείται ο Άγιος των Τελωνιακών ε, και γι' αυτό το λόγο κάνω μια μικρή στάση εδώ στην ιστορία. Λοιπόν, ελληνορωμαϊκός κόσμος, επανέρχομαι, έρεαν οι εμπορικές συναλλαγές, ήταν οι ήπιοι φόροι, οι ήπιοι δασμοί, ανθούσε το εμπόριο σε πάρα πολλές περιοχές και αν ανατρέξουμε ή ε, περάσουμε αν θέλετε αντίστροφα στο μεσαίωνα μετά από χίλια χρόνια τροποποιείται άρδιν το τοπίο. Δεν υπήρχε εμπόριο, κανένας δασμός, κανένας φόρος διότι τότε δεν ενδιαφερόταν ε, για να οικοδομήσει νεόδικα δίκτυα, για να προωθήσει τις εμπορικές συναλλαγές κτλ. Αφετέρου τελωνιακοί σταθμοί και αποθήκες ε, ε, παρέμειναν όταν υπήρχαν και χρησιμοποιήθηκαν για να εκβιάζονται χρηματικά ποσά από τους ταξιδιώτες. Αλλά δεν είχαν συγκεκριμένο στόχο να λειτουργούν στα πλαίσια μιας υγιού οικονομία. Κατόπιν έρχεται και ο προστατευτισμός ε, με την πιο σύγχρονη εποχή. Ε, αλλά ο στόχος δεν ήταν να ισχυθεί το εμπόριο. Το θέμα ήταν να ο, ε, ορθώσει κάθε χώρα φραγμούς για να προστατευτεί από τις γειτονικές χώρες. Και μετά Έχουμε την ε, στροφή ε, στις αρχές του 19ου αιώνα 180 ε, μοίρων γιατί όλοι οι τεχνίτες που αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση οι χώρες χαμήλωσαν τους φορολογικούς φραγμούς τα φορολογικά τείχη που είχαν ορθώσει μειώθηκαν οι δασμοί και σε τέτοιο επίπεδο ορισμένες φορές που δεν υπήρχαν φόροι, δεν υπήρχαν τέλη για κάποια προϊόντα ε, και αυτό που είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το εξή. Ε, βλέπουμε ε, την εθνική ενοποίηση, το κίνημα στη Γερμανία και στην Ιταλία που συνοδεύτηκε από τη εξελίξεις στον χώρο των τελωνίων. Τότε υπήρχαν πολλά μικρά κρατήδια και στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, έπρεπε κάποια στιγμή να καταργηθούν οι δασμολογικοί φραγμοί για να δημιουργηθεί η νέα Γερμανία και να εφαρμόσει ένα ενιαίο δασμό ε, προ τα έξω. Αυτό ήταν το πρώτο μοντέλο, αν θέλετε. Και μετά ακολούθησε το μοντέλο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το ίδιο έγινε ε, και ζητήθηκε να γίνει το ίδιο πάλι με τους δασμούς ε, και να εφαρμοστεί ένας ενίος δασμός ε, προς τα έξω. Ε, ίσως έχουμε ξεχάσει το εξής. Τα τελωνία κατάφεραν να εξυγχρονιστούν 1,5 χρόνο νωρίτερα. οπότε μπορεί κανείς να πει ότι πρώτη φορά στην ιστορία κατάφερε μια υπηρεσία να ολοκληρώσει το έργο τη ένα χρόνο, μισή χρόνο πριν το προβλεπόμενο. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, the... Συνεχίστηκε όμω η ιστορία και μετά τον κοινό δασμό προέκυψε και μια άλλη ανάγκη να ολοκληρωθεί η εναρμόνιση των τελωνιακών διασαφήσεων. Αυτό ε, άργησε πολύ περισσότερο, δεν ολοκληρώθηκε πριν το 1992 αλλά και δεν σήμανε και το, το τέλος των εξελίξεων. Στη δεκαετία του 80 ξαφνικά τα, μειώθηκαν τα εισοδήματα από τα, τα τελωνιακά εισοδήματα. Είχαμε το κίνημα του Γκάτς για τη μείωση ε, των δασμών και οποιονδήποτε άλλων ε, φραγμών ε, στο εμπόριο. Είχαμε μειωμένα λοιπόν τέλη, αλλά τελικά δεν έπεσαν έξω τα τελωνία, απλώς ανέλαβαν ένα νέο έργο. Ε, είχαμε νέες απειλές ε, από το εξωτερικό, όπως αντιλαμβανόντουσαν τουλάχιστον τις εξελίξεις ε, τα, τα κάποια κράτη ως απειλές και άρα χρησιμοποιούσαν τα τελωνία για να ασχοληθούν με θέματα ασφάλειας παραδείγματος χάρη και ανέκυψαν περιορισμοί απαγορεύσεις έφνης που ανέλαβαν οι τελωνιακές αρχές. Αυτή ήταν η πρώτη τελευταία εξέλιξη. Μετά έχουμε και μία τελευταία πριν από μία δεκαετία είχαμε την 11η ε, Σεπτεμβρίου με τις ε, αστυνομικές ε, και αντιτρομοκρατικές δυνάμεις που δεν είναι οι πρώτες που αντέδρασαν, οι τελωνιακές αρχές αντέδρασαν πρώτες διότι έπρεπε να αντιδράσουν σε σχέση με κάποιο κίνδυνο που ε, ε, σχετίζεται με τη μεταφορά εμπορευμάτων. Ε, και μπορείτε να δείτε ότι έχουν γίνει πολλές σοβαρές προσπάθειες για την τροποποίηση του σχετικού κανονισμού το 2005 και τώρα περατώναν τις τελευταίες λεπτομέρειες αναθεώρησης του κανονισμού περί ασφαλείας. Περνάμε στην τελευταία διαφάνεια. Κανονικά θα, θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα έχουν μια νέα καθιερωμένη θέση στα τελωνία πια, αλλά δεν ισχύει αυτό. Ε, πριν από ένα εξάμεινο μπορεί να ακούσατε ότι ε, υπήρχε ε, ένα θέμα με ε, παγιδευμένο δέμα που εστάλει από την Ιεμένη προς τη ΣΥΠΑ και συνειδητοποίησαν όλοι ότι η Τρομοκρατικέ απειλέ ε, δεν ερεμπαίνουν στη ΣΥΠΑ ή στην ΕΕ ε, μέσω ανθρώπων που ταξιδεύουν αλλά και μέσω εμπορευμάτων. Ε, εμείς γνωρίζουμε αυτό το κίνδυνο αλλά όχι απαραίτητα το ευρύτερο κοινό και δεν είχε ασχοληθεί τα μέσα μαζική ενημέρωση με το θέμα της ασφάλειας ε, ε, στα ταχυδρομικά δέματα. Αυτό έγινε το 2010, μία βόμβα που προερχόταν από την Ιεμένη, πέρασε μέσα από τη Γερμανία ε, και σταμάτησαν το παγιδευμένο δέμα στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά όχι επειδή υπήρχε ε, κάποιος ε, έλεγχος ρουτίνας, υπήρχε κάποιο σύστημα ελέγχου Απλώ υπήρξε κάποιο αποτελεσματικός πληροφοριόδότη στον αραβικό κόσμο. Ε, δεν ε, ε, υπήρχε κάποιο σύστημα δηλαδή. Έτσι αποσοβήθηκε η κρίση. Αυτό που με ξαφνιάζει και το ίδιο και κάποιο άλλο είμαι σίγουρο είναι το εξή, ότι στα ΜΜΕ δεν ακούστηκαν οι Υπουργοί Οικονομικών που εκπροσωπούν και τα τελωνία τρόπον αλλά είχαμε στη Γερμανία τον κύριο Ντελεμαζιέρ, τον Υπουργό Εσωτερικών. Ε, ο Υπουργό Μεταφορών επίση, συζητούσε μαζί του σχετικά με τον σχεδιασμό ενός νέου συστήματο κατά αυτή τη απειλή λόγω τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Δεν Κανένας από τι ε, τελωνιακέ αρχές ε, δεν εκλείθη να τοποθετηθεί. Μας ενημέρωσαν απλώ από το ε, Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν βρήκαν ότι θα ήταν χρήσιμο να τοποθετηθούμε κι εμεί. Βλέπετε ότι το κοινό δεν είναι και σίγουρο ποιο διαχειρίζεται τους κινδύνου που σχετίζονται με την αποστολή δεμάτων. Καλό θα ήταν ίσω να καταδείξουν τα τελωνία τι έχουν καταφέρει από το 2005 και μετά και τι μπορούν να καταφέρουν στο μέλλον. Την περασμένη εβδομάδα ε, είδα εδώ στις Βρυξέλλες ένα έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η κυρία Μάλμστρομ, ο κύριος Κάλλας και ο κύριος Εμέτα, τρεις επίτροποι, συνέταξαν από κοινού μια επιστολή ε, σχετικά με το ε, Πώ θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση κατά την άποψή του με ποια νέα συστήματα κτλ. Αλλά και πάλι εδώ οι τελωνιακέ μέθοδοι, οι ρυθμίσει δεν ήταν στην πρώτη γραμμή. Ε, φαινόταν όλα να συμβαίνουν στο Συμβούλιο των ε, Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μεταφορών. Καμία σχέση με τα τελωνία πάντως. Θέλω να κάνω αυτή την παρατήρηση γιατί ίσως αυτό θα εξηγήσει και πολλά στοιχεία που θα μας απασχολήσουν στη σημερινή συζήτηση. Κάτι άλλο τώρα ε, που δεν σχετίζεται με την πολιτική των ΜΜΕ. Ήθελα να μιλήσω για την νομοθεσία. Βρήκα ότι έγινε μια αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση ως προς την έννοια της ε, διαχείρισης ε, των συνόρων και πώς εξελίχθηκε αυτό το σύστημα από το 2001 μέχρι τούδε. Ε, Υπήρξαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΛΑΚΕΝ ναι, το 2001, αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, όπου αναφέρεται μια νέα προσέγγιση για την ε, συνοριακή διαχείριση, δηλαδή μια ευρία έννοια, όπου κάθε αρχή που εμπλέκεται με τη διαχείριση των συνόρων οφείλει να συμμετάσχει. Κυρίως οι συνοριοφύλακες και οι αστυνομικές και τελωνιακές ε, ε, αρχές. Λίγα χρόνια μετά, στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων το Δεκέμβριο του 2006 ε, στα συμπεράσματα ε, υπήρχε ένας ορισμός σχετικά με το, την ολοκληρωμένη συνοριακή διαχείριση αλλά ήταν πολύ στενότερη η έννοια, δεν είχε σχέση με την ασφάλεια ε, περιοριζόταν κατά το μάλλον το ήτον στα αστυνομικά ζητήματα και στους συνοριαφύλακες και στα τελωνιακά ζητήματα και έκτοτε ακολουθούμε αυτή τη γραμμή. Τώρα, στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, για την ε, πολιτική εξωτερικής ασφάλειας ε, έχει εκπονηθεί ένα άλλο έγγραφο που έρχεται να προσθεθεί σε όλα τα υπόλοιπα που προσπαθούν να πλαισιώσουν την εξωτερική μας πολιτική. Επίσης, θέλω να σας πω το εξής. Επιβεβαιώθηκε το δικό μας όραμα, δηλαδή η συνοριακή διαχειρίσει είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του κεφαλαίου 5 για τη δημιουργία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Εκεί μιλάμε για ελέγχους ε, που σχετίζονται με ε, ανθρώπους. Ε, όχι, δεν μιλάμε για έλεγχο εμπορευμάτων, δεμάτων κτλ. Και γιατί το λέω αυτό. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια παρανόηση ως προς τη διαχείριση των συνόρων ότι θεωρείται ευρέως ότι είναι θέμα ασφάλειας, θέμα αστυνομικών δυνάμεων αλλά όχι τελωνιακών ε, αρχών. Ας επισπεύσουμε λίγο Προχωρώντα στην επόμενη διαφάνεια, με αυτή την εισαγωγική παρουσίαση νομίζω σα τοποθέτησα σε σχέση με την κατάσταση όπω έχει τώρα και θα ήταν σκόπιμο να δείτε ε, ποιες, ποιο είναι το δυναμικό, ποια είναι η ικανότητα των τελωνίων ε, τη σήμερα ημέρα και ίσω να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε για ποιο λόγο διαμορφώθηκε όπω διαμορφώθηκε η κατάσταση και τι μπορούμε να κάνουμε. Βλέπετε ότι απαριθμώ διάφορα στοιχεία εδώ. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, τα βλέπετε και στη διαφάνεια. Ορισμένε φορές πάντως υπάρχουν ε, αντικρουόμενες αρμοδιότητες και υπάρχουν παρανοήσεις σε σχέση ε, με ε, τις αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να είχαν τελωνιακές αρχές σε αυτό το θέμα. Ορισμένες φορές προτιμούν τα τελωνία να εισέλθουν στη χώρα τα εμπορεύματα και εκεί να κάνουν τον έλεγχο και όχι στα σύνορα, αλλά Ε, σε σχέση με την πολιτική διαχείριση του κινδύνου θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε ένα νέο σύστημα ούτως ώστε να δραστηριοποιούνται στα σύνορα ε, οι τελωνιακές δυνάμεις ε, όταν χρειάζεται. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Υπάρχουν ορισμένε φορέ δυσκολίες. Δεν είναι θέμα αποτελεσματικότητας Πρόκειται για ένα αντικειμενικό γεωγραφικής φύσεως πρόβλημα που εμποδίζει ορισμένες φορές την ε, διυπηρεσιακή συνεργασία. Διαφέρουν τα σύνορα, ανάλογα αν μιλάμε για χερσαία σέγγεν σύνορα, ε, για θαλάσσια σύνορα. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές ανάλογα με τον τύπο σύνορων, οπότε μόνο 45% ε, των σύνορων ελέγχονται και από τους νοριοφύλακες και από τις τελωνιακές ε, αρχές ε, και άρα ε, ίσως υπάρχει, δεν υπάρχει μεγάλη προθυμία για συνεργασία. Κάτι άλλο από πλευρά μας, ε, ε, ομοιόμορφη εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων. Το τελωνιακό δίκαιο είναι ένα ε, ε νομοθετικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωση που πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά λόγω παραδόσεων, εθνικών παραδόσεων δημιουργείται μια διάσταση απόψεων σχετικά με την ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Θα έπρεπε λοιπόν να τίνουμε όλοι προς την ε, ομοιογενοποίηση των εφαρμοστικών διατάξεων. Αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει να το ρυθμίσουμε εν ώψη και του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα που εμπεριέχει κάποιες ε, πολλά υποσχόμενες ρήτρες προς αυτή την κατεύθυνση και ε, σχέδια. Από θα μας απασχολήσει αυτό το ζήτημα. Επόμενη διαφάνεια. Έχουμε και άλλα, άλλες ελλείψεις ε, οι κυρώσει, τελωνιακέ κυρώσει που ήδη προβλέπονται και άλλου τρόπου για να επιτύχουμε αυτή την ομοιομορφία που επιζητούμε, για την οποία σα έλεγα προηγουμένω. Οι κυρώσει δεν είναι ο μόνο τρόπο. Επίσης ε, μιλάμε για διοικητικές ε, κυρώσει, και, αλλά και κυρώσει ποινικού δικαίου. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η ομοιομορφοποίηση των διατάξεων αυτών και μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας δυσχεραίνουν τα πράγματα. Δεν φαίνεται ότι θα συμβούν σύντομα όλα αυτά. Πάντως θα μπορούσαμε να βρούμε άλλους τρόπους ώστε να είναι ομοιόμορφο το καθεστώς που εφαρμόζεται από όλα, όλες τις τελωνιακές αρχές. Πάντως ο εξυγχρονισμένος τελωνιακός κώδικας και τα νέα τελωνία που θα αρχίσουν να ισχύουν από το 2013 και μετά προβλέπουν ότι θα ε, εφαρμόζονται ομοιόμορφες διατάξεις από όλες τις διοικήσεις ε, παρότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν 27 διαφορετικά, συγγνώμη, διαφορετικές τελωνιακές αρχές ε, θα υπάρξει ομοιόμορφη εφαρμογή. Θα δούμε. Σε σχέση με τη δεκαετία του 80 και του 90 θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει και πολύ μικρότερη χρηματοδότηση για τα τελωνία. Πολλά προγράμματα στην εποχή της ενιαίας αγοράς διοχέτευαν ψηλά κονδύλια για τη, προς τα τελωνία το δεν συμβαίνει πια και υπάρχουν μεγάλε αποκλήσει σε σχέση με το χώρο Σέγγεν. Στο χώρο Σέγγεν υπάρχουν πολλά κονδύλια ε, για τα σύνορα μεταξύ άλλων. Μπορούν να έχουν πιο σύγχρονο εξοπλισμό, να κάνουν νέα προγράμματα κατάρτιση κτλ. κτλ αλλά τα γνωρίζετε αυτά. Τώρα, πολιτική υποστήριξη, όπω σα έλεγα και προηγουμένω, είναι ένα πρόβλημα ε, του Υπουργού Οικονομικών που μεταξύ άλλων είναι αρμόδιος και για τα τελωνία. Και ακριβώ επειδή είναι αρμόδιο για τόσα πολλά ζητήματα, δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τα τελωνία όσο για τον προηγούμενο προπολογισμό. Τώρα ο Υπουργό ε, Εσωτερικών θα ασχοληθεί με του συνοριοφύλακε. Αυτή είναι η ναυαρχίδα του. Δεν πρόκειται να διοχετεύσει κονδύλια για κάτι άλλο. Ε, για θα θέλει να ευχαριστήσει αυτού που τον βγάζουν. Οπότε θα περάσω τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Τη δεκαετία του 90 είχαμε ε, ένα απλό τοπίο, μία γάμα δέλτα, Γενική Διεύθυνση και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γάμα δέλτα 21 τη λέγανε, η ταξούντ δηλαδή η σημερινή που ε, κάλυπτε όλες τις πιθανές λειτουργίες των τελωνίων. Και τώρα το 2010 έχετε καταμερισμό όλων των αρμεδιοτήτων σε διάφορες υπηρεσίες. Ταξούντ, Όλαφ, DG Εσωτερικών Υποθέσεων, ε, Ομάδα Εργασίας ε, για την Τελωνιακή Συνεργασία του Συμβουλίου και το καθεξής. Οπότε δεν συνιστούν όλοι αυτοί έναν ενίο συνομιλητή ενώπιον της Frontex αν θέλουμε να επικρατήσει μεγαλύτερη συνοχή στη διαχείριση των συνόρων μας. Επόμενη διαφάνεια, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, ε, όμως ε, βλέπετε σαφέστατα πως τα διάφορα ε, μοντέλα που έχουμε για την ολοκληρωμένη συνοριακή διαχείριση ε, μεταξύ αυτών έχουμε ένα που αποφάσισε το Συμβούλιο το 2006 όπου έχουμε ένα πολύ στενό ορισμό που όμως δεν μας βοηθάει διότι εστιαζόμαστε στα θέματα ασφάλειας και τα αστυνομικά ζητήματα. Χρειαζόμαστε μια ευρύτερη διεθνή έννοια που χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Ένωση Τελωνίων και ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενστερνιστεί αυτή την ε, έννοια που χρησιμοποιεί στις σχέσεις τη με τρίτε χώρες. Δεν εφαρμόζεται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Ο στόχος μας, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι να εφαρμόσουμε αυτή την ευρύτερη διεθνή έννοια γενικότερα, γιατί εμπλέκονται όλες οι υπηρεσίες, όλοι οι οργανισμοί που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η ασφάλεια ότι όλοι ό,τι σχετίζεται με τη διαχείριση των συνόρων θα λειτουργεί κάτω από την ίδια ομπρέλα αν θέλετε. Επόμενη διαφάνεια. Τι μπορούμε να προβλέψουμε μελλοντικά για τα τελωνία. ούτω ώστε να υπάρχει ένας ε, ομότιμος, ένας συνομιλητής ε, για τον Frontex ε, θα μπορούσαμε να έχουμε μια αυτοτελή υπηρεσία τελωνίων. Έχουμε την ECA, European Customs Agency, ε, το πρόβλημα είναι ότι ή είναι πρόβλημα χρηματοδότησης, δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια ή δεν επαρκεί ένας οργανισμός ε, για να συντονίσει όλες αυτές τις δράσεις. Όμως αλλάζουν οι απόψεις κοινοτροπίες. οι ε, Κάποιοι θεωρούν ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο χρειάζεται συντονισμός ανάμεσα στους οργανισμούς που ασχολούνται με την συνοριακή διαχείριση, άλλους που ασχολούνται με την ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου κτλ. κτλ. Ε, θα μπορούσε λοιπόν ένας τέτοιος νέος οργανισμός να συμβάλλει και σίγουρα θα είναι αποδοτική η επένδυση αν αποφασιστεί να συσταθεί ο οργανισμός. Άλλες εναλλακτικέ λύσεις που συζητούνται είναι η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα τελωνιακά ζητήματα να αναλάβει αυτό το ρόλο. Αυτό δεν είναι καλή ιδέα γιατί δεν έχουν υποδομή, δεν έχουν εξοπλισμό, εξαρτώνται από την εκάστοτε προεδρία, οπότε πώς να αναπτυχθεί ε, μια ολοκληρωμένη και συνεκτική ε, προσέγγιση. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε μια υπηρεσία τελωνίων στο εσωτερικό των υφισταμένων οργανισμών χρηματοδοτικούς, πώς είναι πιο ενδιαφέρον αυτό, αλλά τα τελωνία θεωρούν ότι ε, θα είναι κακό για την εικόνα των ε, τελωνίων ε, είτε μιλήσουμε για υποτμήμα της Europol είτε του Frontex. Δηλαδή δεν θα βοηθούσε αυτό την εικόνα των τελωνίων. Πώς θα εξηγήσουν τα τελωνία στο ευρύτερο κοινό το ρόλο τους αν γίνει αυτό. Θα χάσουν κάθε προβολή. Τώρα αυτός ο αυτοτελής οργανισμός, η πρώτη λύση που σχολίασα, μπορούν να συμμετάσχουν όλοι η Όλαφ ε, συνδέεται στενά με τα τελωνιακά ζητήματα ε, γιατί προέρχεται από την παλιά Γενική Διεύθυνση 21 και είναι ισχυρή ακόμη η δεσμή αλλά φυσικά δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε εδώ αυτό. Θα το συζητήσουμε λεπτομερέστερα. Θα ήθελα να ε, σχολιάσω επίσης σε κάποιες απόψεις όπως αυτή των Γάλλων που θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να γίνει μια μελέτη πριν συσταθεί ο οργανισμός ε, ECA, αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Τελωνία. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι υποσυζήτηση διάφορες ε, ιδέες. Περνώ στην τελευταία διαφάνεια για να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου. Ε, φυσικά υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων στην Ευρώπη για το θέμα. Ελπίζω να υπάρξει συντονισμός και να ολοκληρωθούν ναι, υπό μια ενιαία αιγίδα όλα τα ζητήματα, όχι απαραίτητα όπως τη είπα να υπάρχει μο, ε, μια συνοριακή υπηρεσία όπου συλλειτουργούν ε, τα τελωνία ε, και η αστυνομία. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε υπό κάποια άλλη μορφή, μέσω ενός δικτύου. Αυτή ήταν και η πεμπτουσία της παρουσίασής μου, αυτή η τελευταία μου πρόταση. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ και α, ε, μας δώσατε αρκετά ερεθίσματα. Προφανώς ε, κάποια ζητήματα δεν είναι άμεσης αρμοδιότητας της Επιτροπής μας, αλλά νομίζω πως η έκκλησή σας για καλύτερο συντονισμό πράγματι είναι πολύ σωστή και ξέρουμε πως θα έχουμε σύντομα μια νομοθετική πρόταση περί εφαρμογής ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τα τελωνία και βλέπετε πόσα πράγματα φορτώνονται ήδη στα τελωνία πέρα από τον ρόλο του προστασίας των εισοδημάτων του κράτους όπως είπατε και στην ιστορική σας αναδρομή. Λοιπόν, έχουμε αρκετό χρόνο για ερωτήσεις. Να σας υπενθυμίσω πως ε, δεν κάνουμε ανταλλαγές απόψεων για την έκθεση Σαββίνη, απλά για να δούμε το τι γίνεται με την έκθεση Επιτροπής ε, Ελευθεριών. Και χαιρόμαστε που είστε εδώ πέρα παρά το ότι δεν ε, βρήκαν τον ανάλογο χρόνο στην συνάδελφοι της Επιτροπής Ελευθεριών. Ποιος θα να ξεκινήσει, κυρία Τούν? Κάνουμε ένα γύρο από όσοι προσωπούν τους, τους σκιώδους. Ε, να μιλήσω εξ ονόματος ε, του σκιώδου ή εξ ονόματος μου. Πρώτα εξ ονόματος σκιώδους. Γιατί είναι διαφορετικά τα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει. Ο πρόεδρος, ξεκάθαρα πως δεν, είπα ξεκάθαρα πως δεν θα συζητήσουμε την έκθεση Σαββίνη σήμερα. με βάση αυτά τα οποία μας είπε ο συγητή μα. Μάλιστα, η κυρία Κοριόλα η οποία λείπει μου είπε πως ε, κοίταξε τη μελέτη σα. και επειδή βεβαίω ε, δεν μπορεί να παραστεί μου ζήτησε να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτή και αυτό το οποίο τονίζει είναι πως Βλέπουμε σαφώς πως χρειάζεται συντονισμός σε τελωνιακά ζητήματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα τομέα που δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου συντονισμός αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές στα εξωτερικά μας σύνορα αυτή τη στιγμή η διαχείριση από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μειωμένη μόνο μεταξύ αστυνομικών αρχών υπό τον συντονισμό της Frontex χωρίς εμπλοκή των τελωνίων. Όπως είπατε στη μελέτη, ο αποκλεισμός των τελωνίων από τη διαχείριση των συνόρων ε, δεν ε, συμφωνεί με διεθνείς προδιαγραφές. Στη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας αναφέραμε το ζήτημα των ηλεκτρονικών τελωνίων και πόσος χρόνος χρειάζεται πραγματικά για να είναι έτοιμο το σύστημα πληροφορικής ε, υπομορφή που απαιτεί ο εξυγχρονισμένος ελληνιακός κώδικας. Κάποιοι λένε πως μπορεί να γίνει σύντομα, ακόμα και μέχρι το 2013. Και η συναδελφός μου, κυρία Κορολα, θα ήθελε την άποψή σας και το τι θεωρείτε εσείς ως κίνδυνο αν επιμείνουμε στην αρχική προθεσμία του 2013 και ε, τι θα γίνει αν ε, δώσουμε περισσότερο χρόνο. Ένα άλλο θέμα, λέει η συνάδελφος, είναι πως ε, εξετάζεται τις αρμοδιότητες και δυνατότητες των τελωνίων και έχουμε δει το ζήτημα της εποπτείας αγοράς ε, στην Επιτροπή μας νωρίτερα φέτος και καταλήξαμε στο ότι η συνεργασία τελωνίων με τις αρχές εποπτείας αγοράς πρέπει να προχωρήσει. Και το ερώτημά της είναι τι θεωρείτε εσείς ότι είναι τα υπέρ και τα κατά της στενότερης συνεργασίας μεταξύ ε, τελωνιακών αρχών και αρχών εποπτείας της αγοράς και τέλος μου ζήτησε να σας πω το εξής τις ΕΠΑ έχουν τις απαιτήσει ε, σάρωσης 100% των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα ε, βεβαίως απέχουμε από αυτό τελείως συμπτωματικά εγώ ήρθα α, μέσω, έφερα μέσω Στρασβούργου και Βαρσοβίας και Φραγκφούρτης ένα μαχαίρι στη βαλίτσα μου το οποίο το ανακάλυψα στη Βαρσοβία ε, κάπου τόσο και πέρασε από όλες αυτές τις μηχανές οπότε κατά την άποψή σας ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε περισσότερη σάρωση ή καλύτερη αξιολόγηση κινδύνου. Αλλά βρήκαν δύο καρότα στην ίδια βαλίτσα και τα μελέτησαν πολύ προσεκτικά. Αλλά άφησαν το μαχαίρι. This was last week. <laughs> Την προηγούμενη εβδομάδα όλα αυτά που σας λέω. Έχω και φωτογραφία του μαχαιριού, εάν σας ενδιαφέρει, γιατί ήταν πολύ συναρπαστικό όταν το βρήκα στη χειραποσκευή μου όταν προσγειώθηκα και το έβγαλα φωτογραφία. Σας ευχαριστούμε για αυτές τις αποκαλύψεις. Ε, είχατε το μαχαίρι για να καθαρίσετε τα καρότα, ίσως. Εν κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ και εγώ το ίδιο σκέφτηκα. Και εγώ σκεφτόμουν το ίδιο για το μαχαίρι και τα καρότα, αλλά τέλο πάντων, πέρα των αστυνομών, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον παρουσιαστή για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση που δείχνει επίση ποιοι σύνδεσμοι υπάρχουν μεταξύ των επιτροπών. Και νομίζω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Ήθελα να θέσω μια πληρώτηση για τους σπόρους. Ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, με τις δημόσιες περικοπές, στις περικοπές του δημοσίου τομέα, σε πολλές αυτές τις υπηρεσίες ε, που μας προστατεύουν, αντιμετωπίζουν ε, θέματα δημοσιονομικού χαρακτήρα, τέτοιου είδου προβλήματα. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω, αναφερθήκατε στο θέμα της συνεργασίας, στη δικτύωση που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Υπάρχει ένας τρόπος να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τους πόρους για την ασφάλεια, αλλά έχετε σκεφτεί για κάτι σε σχέση με τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει κάτι τέτοιο στην ασφάλεια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και το θέσατε πάρα πολύ εύλογα το παράδειγμα της Ιεμένης ε, ήταν ε, μάλλον ε, στρατηγικές πληροφορίες, μυστικές πληροφορίες που δόθηκαν εκεί. Αλλά θέλω να ρωτήσω και για τη Frontex. Πώς βλέπετε τη συνεργασία, νομίζω και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά καθώς μιλάμε για την τελωνία και την μεταρρύθμιση και το θέμα του χρονοδιαγράμματος, αναφερθήκατε και σε ζητήματα τεχνολογίας των πληροφοριών. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να τα εξετάσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα, γιατί όλους μας ενδιαφέρει η ασφάλεια και η αποδοτικότητα, αλλά και το πώς χρησιμοποιούμε τους πόρους. Ευχαριστώ. Uh, euh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι δύσκολο εδώ πέρα να ξεχωρίσουμε τη συζήτηση εσωτερικής αγοράς από την έκθεση στην Επιτροπή Ελευθεριών, αλλά θα προσπαθήσω να μείνω εντός του πλαισίου εμείς ε, βεβαίως ξέρουμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικά τα τελωνία για την εσωτερική αγορά, ο έλεγχος π.χ. μαϊμούδων, προϊόντων απομιμήσεων, αλλά αυτό το οποίο είναι επίσης σημαντικό και το είδαμε και στην ε, ε, παρουσίαση είναι ή διαφορετικές ε, συνθήκες που αντιμετωπίζουν ε, ε, π.χ. οι επιβάτες στα αεροδρόμια όπως ακούσαμε, π.χ. εντός της ζώνης έγκαινο που δεν υπάρχει ενεργητικός έλεγχος και δεν είναι σαφές νομίζω το τι γίνεται και θα έπρεπε ίσως να υπάρχει μια διαφώτιση του Ευρωπαίου πολίτη για το τι κάνουν τα τελωνία και τη διαφορά μεταξύ Σέγγεν και Τελωνιακής Ένωσης. Και το ότι αυτό το οποίο μας φαίνεται ως ενδοευρωπαϊκό σύνορο μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικά καθεστώτα. Έχω κάποιες ε, παρατηρήσεις για κάποια κένα κατά την απόψή μου που θα ήθελα να συμπληρωθούν. Βλέπουμε εδώ πέρα στην παρουσίαση πως ε, γίνονται πάρα πολλά για τα χερσαία σύνορα, αλλά ξέρετε πως στην Ολλανδία έχουμε και αεροδρόμια και λιμάνια και δεν ε, μας είπατε πάρα πολλά σχετικά. Να δούμε επίσης τι γίνεται με την ε, τεχνολογία. Μας είπατε για τον αυτοματισμό, αλλά στα θαλάσσια λιμάνια, ξέρετε στο Ρότερνταμ, έχουμε αυτές τις συσκευές ε, σάρωσης, αλλά δεν ισχύει το ίδιο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντικό είναι να δούμε και τις ε, τεχνικές που υπάρχουν εκεί πέρα και τυχόν εισαγωγή τέτοιων ε, τεχνολογιών. Αυτό το οποίο επίσης δεν άκουσα στην έκθεση που είναι ισιώδες ε, νομίζω είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς. Ε, ε, καλοί κανόνες και οι ποινές, ωραία όλα αυτά, αλλά το πώς εφαρμόζονται έχει μεγάλη σημασία και βέβαια είναι κλειδί για τα τελωνία ή η διαφθορά και είναι κάτι το διεθνές ε, βεβαίως και νομίζω πως θα έπρεπε να αναφερθεί στην παρουσίαση Και τέλος οι λύσεις. Ε, υπηρεσίες τώρα, άλλη μια υπηρεσία δεν θεωρώ πως χρειάζεται. Έχουμε πάρα πολλές ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα μια πρακτική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και σε συνδυασμό με αστυνομία και άλλες ε, υπηρεσίες ε, για να έχουμε μια νέα μορφή συνεργασίας. Αυτό το οποίο δεν είδα όμως την παρουσίαση σας είναι η συνεργασία στον Παγκόσμιο Τελωνιακό Οργανισμό που είναι πράγματι έντονη. Έχω πάει σε τέτοιες ε, συνεδριάσεις αυτού του οργανισμού. Είναι πάρα πολύ πρακτικά τα ζητήματα και οι συζητήσεις που γίνονται και νομίζω θα έπρεπε και αυτό να το λάβετε υπόψη. Ευχαριστώ κύριε Ράπτη. Κάποιος άλλος και ο κύριος Σμιτ. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα προηγουμένως την περιπέτεια που είχε η Ρόζα με το μαχαίρι και το καρότο και σκέφτηκα ότι ε, συνήθως λέμε για μαστίγιο και καρότο η Ρόζα τώρα μας έβαλε σε ένα άλλο, σε μια άλλη ιστορία μαχαίρι και καρότο. Ε, είναι από αυτά τα διάφορα που συμβαίνουν ε, και σκέφτομαι το εξής. Έλεγχος. Ε, κάποιος μπορεί να περάσει ένα μαχαίρι ή ένα καρότο. Επειδή εγώ προέρχομαι από την Ελλάδα και έχουμε όπως και ο κύριος De ε, πολύ πολλή θάλασσα γύρω μας ε, και αεροδρόμια και λιμάνια και χερσαία σύνορα και έγινε αναφορά και στη Frontex ε, υπάρχουν περιπτώσεις εκτός από μαχαίρια και καρότα να περνάνε άνθρωποι λαθρομετανάστες κρυμμένοι μέσα σε φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα. Βάζω μια άλλη διάσταση που εκ των πραγμάτων περνάει ε, ε, μια νταλίκα, ένα πολύ μεγάλο φορτηγό που φεύγει για παράδειγμα από την Πάτρα ή που μπαίνει στην Πάτρα, ε, περνάει έλεγχο. Στον έλεγχο δεν είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν όλα όσα περιέχει μέσα το φορτηγό ένα παράδειγμα. Ε, πρέπει να το δούμε και αυτό λίγο. Ε, και το άλλο θέμα που θέλω να ρωτήσω είναι το θέμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, πέρα από τους σπόρους που αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Οι άνθρωποι που είναι στα τελωνία, ε, όταν μάλιστα βρισκόμαστε μπροστά στην διαδικασία εξυγχρονισμού των τελωνίων, είναι ένα θέμα που το συζητάμε όπως ξέρετε στην επιτροπή μας ε, υπάρχει το θέμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης της προσαρμογής ε, στις νέες τεχνολογίες. Ε, τέλος κλείνοντας να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης. ήταν πολύ γλαφυρά δοσμένα όλα όσα είπατε ε, ήταν, δεν ήταν μια συνηθισμένη τεχνοκρατική παρουσίαση και αυτό την έκανε να είναι πιο προσιτή όχι μόνο σε εμά που δουλεύουμε για αυτή την υπόθεση αλλά νομίζω και σε έναν απλό Ευρωπαίο πολίτη και έτσι δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό. Ε, και να πω τέλος ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η παρουσίαση όταν μάλιστα στις 16 του μηνός ε, μεθαύριο έχουμε μια ακρόαση για αυτό το θέμα Ευχαριστούμε εσάς αλλά ευχαριστούμε και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ελευθεριών που είχαν την ιδέα για αυτή την έκθεση, την ωφέλεια από την οποία πήραμε εμείς. Κύριο Σμιτ, ευχαριστώ. Δυστυχώ, δεν μπορούσα να σας ακούσω. Έπρεπε να λύσω κάποια άλλα θέματα σε μια άλλη συνεδρίαση, αλλά αφού διάβασα αυτό το έγγραφο και είδα και τι διαφανιέ σα εδώ, θέλω να σας θέσω μια άλλη ερώτηση. Ένα από τα κύριε ζητήματα είναι να ανασταλεί όλη η διαδικασία. Και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σα, Αν το πράξουμε αυτό, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και ο αντίκτυπο τη αναστολή τη ολη διαδικασία. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχει πλειοψηφία σε αυτό τον οίκο, αλλά και αυτή είναι και η άποψη τη Κομισιόν. Και μπορώ να πω ότι είμαι κάπω διστακτικό. αλλά θα ήθελα να ακούσω και εσά. Εδώ αναφέρεται ότι η επικράτεια Σιέγγεν και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το ίδιο. Φυσικά αυτό είναι απόλυτα σωστό. Παίρνω το σχάρι. Εγώ ζω στην Νότια Σουηδία και καθημερινά υπάρχει ε, μέσω του ΣΥΠΟΛ υπάρχουν ε, τόνοι το ΚΑΤ ε, και είναι παράνομο στη Σουηδία και καθημερινά το βρίσκουμε, το κατάσχουμε αυτό το υλικό, αυτό το νοικοτικό και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τους ίδιους κανόνες σε όλη την Ευρώπη για το ότι είναι παράνομο. και σε σχέση και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Αλλά σε, η ερώτησή μου αφορά τη ΣΕΝΚΕΝ και την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ε, γνωρίζουμε τώρα ποια είναι η Σέγγεν ε, και ε, υπάρχουν και θέματα με τα σύνορα, είναι υποεπίθεση. Έτσι λοιπόν πώς αυτά τα δύο ζητήματα σχετίζονται μεταξύ τους. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Και τι συμπεράσματα, σε τι συμπεράσματα καταλήγετε εσείς ε, με αυτό το όλο, όλη η πολιτική αναταρχή σε ό,τι αφορά τη Σέγγεν. Δηλαδή αυτό θα επεκταθεί και στα εξωτερικά σύνορα με γενικότερους όρους. Ίσως ήδη έχει γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί δεν ε, έγιναν αποδεκτές η Ρουμανία και η Βουλγαρία ε, στο χώρο Σέγγεν και υπήρχε ένα θέμα εξωτερικών συνόρων. Good. Um, Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν ο κ. Σιτσκι θέλει να παρέμβει για κάποια ζητήματα, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Με ευνηδιάσατε, γιατί εγώ ήρθα εδώ για να ακούσω τον ε, δ. Χόμπινγκ ε, και φυσικά και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά φυσικά να σας πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τη μελέτη. Υπάρχουν πάρα πολλοί χρήσιμες πληροφορίες σε αυτή. Θα έλεγα ότι επικεντρώνεται πέρα πολύ στις πτυχές της ασφάλειας, ε, αλλά βέβαια εφόσον ζητήθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ε, ίσως ε, είναι και λογικό. Βέβαια τα τελωνία δεν συνιστάνται μόνο στην ασφάλεια και η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική. Είδαμε και την παρουσίαση της ε, σωστής εικόνας ε, μελέτη. Ε, είχαμε μία τροποποίηση του 648, λειτουργεί τώρα στα κρατημέλη, αλλά από τότε έχουν αναλάβει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τα τελωνία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των συνόρων και την πτυχή τη ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ΟΛΑΦ. Ε, έχουμε και ε, μεικτέ συνεδριάσει, όπω σε μέτα. Ε, και δεν βλέπουμε το έλλειμμα συνεργασία με την ΟΛΑΦ, ε, βέβαια. Η άποψή μα ενίοτε διαφέρει γιατί έχουμε και διαφορετικά χαρτοφυλάκια. Είναι λογικό, αλλά καθημερινά συνεργαζόμαστε. Και καθώ έχω το λόγο, θα ήθελα μόνο να πω ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες δεν υπάρχει 100% σκάνινγκ, σάρωση, το ζητούν, αλλά ε, διαφέρει η έννοια, γιατί εμείς κάνουμε τη σάρωση πριν ε, να ε, συσκευαστούν τα αγαθά και σταλούν στι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν σαρώνονται στι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά σε όλε τι χώρε εταίρου. Και φυσικά αυτό δεν μα αρέσει, γιατί έχουμε τεράστιο άχθο για το εμπόριο και πολύ ψηλό κόστο. Θα σταματήσω εδώ, Πρόεδρε. Γιατί αν και θα ήθελα να σχολιάσω κάθε σχόλιο που ακούστηκε, δεν είναι ο ρόλος μου αυτός εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Κάποιες από τις πτυχέ αφορούσαν και τον χρόνο του εναρμονισμένου τελωνιακού κώδικα και ίσως να μην είναι βεβαίως ε, στο πλαίσιο της εντολής του κυρίου Χόμπιν εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε ίσως να το συζητήσουμε όταν έρθει και ο κύριος ε, Σολβίνη εδώ πέρα. Λοιπόν, αν θέλετε να απαντήσετε εντό 6 λεπτών για να ε, σεβαστούμε και το ωράριο. Εάν αργήσετε θα κάνω νόημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ να σχολιάσω. Πράγματι ο κύριος ε, Σενίνσκι έδωσε κάποιες απαντήσεις. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα πολύ σωστά είπε. Σε κάποια ζητήματα πρέπει να πω πως βλέπουμε την ε, διαφορά. Υπήρχε μία μελέτη της Κομισιόν και πράγματι συχνά δίνεται περισσότερο βάρος σε ζητήματα ασφαλείας αλλά αυτό έχει και άλλη μία ε, συνέπεια. Δεν μπορώ να σχολιάσω ζητήματα που αφορούν ε, την Επιτροπή σας ε, όσον αφορά δηλαδή την απόφαση που θα λάβετε να, να αναβάλλετε ή να μην αναβάλλετε. Δεν, δεν γνωρίζω το θέμα. Και επίσης την ηλεκτρονική τελωνιακή περιοχή σε γενικές γραμμές μπορώ να πω πως είναι μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση και θα βοηθήσει οπωσδήποτε να κάνει και τις διαδικασίες απλούστερες. σε ολόκληρη την Ευρώπη με το να έχουμε μια κεντρική εικόνα του τι συμβαίνει σε ολόκληρη την τελωνιακή επικράτεια αυτό είναι μια σωστή προοπτική. Τώρα δεν έχω άποψη για το εάν είναι δυνατόν από το... μέχρι το 2013 γιατί δεν, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες οπότε δεν θα σχολιάσω. Επίσης για την επαφή μεταξύ τελωνιακών αρχών και αρχών εποπτείας αγοράς ακούγεται πολύ θετικό. Και πάντα το να έχουμε περισσότερες ανταλλαγές πληροφοριών είναι καλό αλλά ούτε σε αυτό το θέμα είμαι ειδικό. Αντιθέτως, όσον αφορά την σάρωση 100% στη ΣΥΠΑ, αυτό το θέμα με έχει απασχολήσει και έχω συνεργαστεί με Αμερικανούς ε, ε, υπαλλήλους. Ε, το 100% ήταν πάντα ο επιθυμητός στόχος για τη ΣΥΠΑ ε, επευλήθη από τον ίδιο τον πρόεδρο πως αυτό θα έπρεπε να γίνεται αλλά όταν βλέπουμε τις αναφορές ε, των Αμερικανικών τελωνιακών και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είναι πολύ επιφυλακτική ε, λένε πως δεν είναι δυνατόν υπάρχουν περιπτώσεις οποίες χρειάζεται να ελεγχθεί, να σαρωθεί 100% ενός φορτίου ή επιβατών και δεν, δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο γιατί θεωρώ πως δεν υπάρχει ε, ανάγκη να γίνει τέτοιος έλεγχος. Οπότε υπάρχουν αμφιβολίες και εντός τον είπα για το αν είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο και εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της ιδέας του ότι ένα σωστό σύστημα αξιολόγησης κινδύνου είναι ε, κατά πολύ ανώτερο από μια σάρωση 100%. Και βέβαια σα ευχαριστώ για αυτό το οποίο είπατε για το καρότο και το μαχαίρι. Αυτό συμβαίνει, συμβαίνει και στις είπα. μπορώ να σα πω πολλά τέτοια περιστατικά που ε, λαμβάνουν χώρα στα σύνορα με το Μεξικό για να δείτε τι περνάει εκεί πέρα. Παρά το ότι υποτίθεται πως ε, είναι υποχρεωμένοι να κοιτάνε κάθε αυτοκίνητο και κάθε αποσκευή. Ποτέ δεν είναι πλήρης ο έλεγχος. Οπότε εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, έχω κάποιες επιφυλάξεις. Όσον αφορά τους πόρους, αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, είμαστε πιεσμένοι. Αλλά, εάν τεθεί αυτό νομίζω από πολλά θεσμικά όργανα μπορεί να στείλει ένα πιο ισχυρό μήνυμα. Τώρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση για ε, τα ζητήματα Σέγγεν και ενιαίας αγοράς. Οπωσδήποτε είναι ένα πρόβλημα το ότι έχουμε αυτές τις διαφορετικές επικράτειες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το ότι δεν έχουμε τους ίδιους κανόνες ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα ήταν επιθυμητό, αλλά όπως ξέρετε αυτό είναι ε, ζήτημα πολύ σημαντικό εθνικών προτεραιοτήτων και προτιμήσεων και οπωσδήποτε κάποια κράτη δεν θέλουν να μην έχουν αυτή την αυτονομία και τις εθνικές ε, προτιμήσεις. Αλλά πάλι όταν μιλάμε για έλεγχο σε μια χώρα Σέγγεν πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Το είχαμε εξετάσει αυτό όταν ξεκίνησε η Σέγγεν και όταν ξεκίνησε ακόμα και η ενιαία αγορά υπήρχε πάντα το ερώτημα τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή έχουν καταργηθεί τα σύνορα. Και ήταν πάντα σημαντικό, έχει γραφτεί στη συνθήκη του Μάστριχτ πως ε, τα τελωνία έχουν πάντα την δυνατότητα να κάνουν τους ελέγχους τους και να ελέγξουν ορισμένα φορτία και αυτό ε, μπορεί να γίνει οπουδήποτε στο εσωτερικό της χώρας, σε ένα αυτοκινητόδρομο, στο κέντρο μιας πόλης, στα σύνορα, αλλά δεν θα πρέπει να είναι συστηματική έλεγχη στα σύνορα. Αυτό ισχύει ε, είτε στη ζώνη Σέγγεν είτε όσον αφορά τα τελωνία, ότι δεν θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν ξανά να επιβληθούν ε, μόνιμοι έλεγχοι στα σύνορα. Πρέπει να είναι ad hoc, ε, τυχαίοι και ως ε, πρώην εργαζόμενος στον τομέα της επιβολής το θεωρώ πολύ αποτελεσματικό και αν υπάρχουν έξυπνοι ερευνητές οπωσδήποτε θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως τα αεροδρόμια όπως αναφέρατε είναι κάτι το δύσκολο. Αυτό ισχύει στην Ευρώπη αλλά και στη ΣΥΠΑ πως ε, καμιά φορά ε, οι εσωτερικές με τις εξωτερικές ε, ροές ε, ανακατεύονται και ανακατεύονται φορτία και ταξιδιώτες με διαφορετικούς προορισμούς. Είναι ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν είναι ικανοποιητική οπωσδήποτε κατάσταση, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Για να δω τώρα. Φορτηγά και άνθρωποι που κρύβονται στα φορτηγά και οι τεράστιοι αυτοί σαρωτές, αυτή είναι μια νέα τεχνολογία, όχι τόσο νέα, υπάρχει εδώ και λίγα χρόνια. Αυτό βοηθάει Τώρα, ε, δεν είναι σωστό να αγοράσουν και οι συνοριοφύλακες ε, και τα τελωνία τα ίδια μηχανήματα. Πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός και κοινή χρήση. Και νομίζω μπορεί να γίνουν και οικονομίες κλίμακος. και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Ε, έφτασε στο τέλος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ για τις υποδείξεις σας που θα μας βοηθήσουν ε, με την μελέτη μας και θα ασχοληθούμε και με άλλους ε, τομείς. Εστιάσαμε στους σημαντικούς τομείς η συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών, δηλαδή στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Παγκόσμιος Τελωνιακός Οργανισμός, πάρα πολύ σημαντικός για τις τελωνιακές διοικήσεις, αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα της μελέτης μας. Είναι αυτονόητο πως υπάρχει καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι άξιζε το χειροκρότημα. Και σας καλέσαμε επίσης να έρθετε στην ακρόασή μας, έτσι ώστε οι συνάδελφοι θα έχουν και άλλη ευκαιρία να σας θέσουν ερωτήσεις για αυτές τις πτυχές και νομίζω ότι είναι αύριο, όχι στις 16, την Πέμπτη. Την Πέμπτη έχουμε μία ακρόαση. Έτσι λοιπόν θα τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Να σας υπενθυμίσω ότι η ευρύνη συνεδρία θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί γιατί δεν θα συζητήσουμε το θέμα της καταναλωτικής πίστης, της σχετικής οδηγίας, δεν είναι εδώ εισηγητής, αύριο στις 10 λοιπόν και θα ε, σταλεί σε όλους και κατάλληλη ενημέρωση για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έρθετε στις 9. Έχουμε δύο ψηφοφορίες, ε, καταρχήν για ε, την έκθεση ΒΑΜ και στη συνέχεια έκθεση ΡΕΠΟ και Γκέπχαρτ. Και σας ευχαριστώ όλους. Ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρία. Θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί. Ευχαριστώ.